Νομίζω ότι η τεχνολογία του Skype είναι μαζί μας. Οπότε μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο 10 που είναι η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο Λίβανο. Νομίζω λοιπόν ότι τεχνολογικά είναι όλα εντάξει. Η κατάσταση στο Λίβανο, όπως γνωρίζετε, εδώ και μερικές εβδομάδες έχουμε τον κόσμο στο δρόμο γεωπολιτικά είναι ασταθής η κατάσταση, αλλά υπάρχει και οικονομική και πολιτική κρίση ενδημική. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτήκαμε ότι ήταν σημαντικό να εξετάσουμε τις πρόσφατες εξελίξεις στη χώρα, μια χώρα φίλη, με την οποία έχουμε ιστορικά δεσμούς. Έχουμε ανταλλαγή απόψεων λοιπόν στα πλαίσια ε, το ότι μας ενδιαφέρουν όλα τα κινήματα, τα ειρηνιστικά και οι ειρηνικέ διαμαρτυρίες. Έχουμε κάνει τα ίδια και για την Αλγερία, το Σουδάν και το Χονγκ Κόνγκ. Σήμερα έχουμε δύο εξέχοντες ε, που θα πάρουν το λόγο από την Βηρητό μέσω Skype και θα τους δώσω το λόγο ευθύ αμέσω. Έχουμε τον Καρίμ Ελμουφτή που είναι πολιτολόγος και καθηγητής δικαίου και πολιτικών επιστημών και διευθυντής της νομική κλινική των εισαγωγικών όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Πανεπιστήμιο Σαζέ. Και έχουμε και τον Τζορτζ Γκαλί, που είναι εκτελεστικό διευθυντή τη μη κυβερνητική οργάνωση Αλεφ Αζίρ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δέκα λεπτά παρακαλώ. Έχετε το λόγο, κύριο Μουφτή πρώτα. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα. Ε, ευχαριστούμε που μας ε, δώσατε την ευκαιρία να παρέμβουμε. Ξέρετε ότι έχουμε μία σειρά διαμαρτυριών πρωτοφανή στο Λίβανο. Όχι ότι είναι η πρώτη φορά και η πρώτη φορά που έχουμε ειρηνικές διαμαρτυρίες, αλλά ε, το πρώτη φορά έχει να κάνει με τη μορφή, ότι δεν γίνεται μόνο στη Βηρητό, αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις του Λιβάνου. Και είμαστε στην 16η μέρα κινητοποίησης. Και αυτό στα πλαίσια ε, συσσόρευσης κακών ειδήσεων τα τελευταία χρόνια. Το κοινωνικό και οικονομικό βάρος που επομίζονται οι Λιβανέζοι είναι πολύ μεγάλο και αυτό οδήγησε στο ξέσπασμα των διαμαρτυριών αυτών. Μεταξύ άλλων κακών ειδήσεων μπορούμε να αναφέρουμε ε, την ελευθέρωση των ενοικιών από το 2014, κάτι το οποίο οδήγησε ε, πολλές οικογένειες στην περιφέρεια να αναγκαστούν να φύγουν από τα σπίτια τους. Το θέμα των επιδοτήσεων στη στέγαση μειώθηκε, έπειτα οι φόροι αυξήθηκαν και πιο πρόσφατα έχετε και δύσκολη πρόσβαση σε συνάλλαγμα, σε δολάριο. Και τη 17η Οκτωβρίου είχαμε την περίφημη απόφαση του Υπουργού του Τηλεπικοινωνιών να φορολογήσει το WhatsApp, την εφαρμογή WhatsApp. Οπότε ξέσπασαν διαμαρτυρίες παντού στο Λίβανο. Χάθηκε η εμπιστοσύνη στον κόσμο. Στα πλαίσια αυτά πρέπει να προσθέσω ακόμα <clears throat> και τις ανισότητες στο Λίβανο. Δεν είμαστε οι μόνοι, αλλά υπάρχει τεράστια φτώχεια, μεγάλη διαφθορά, ε, κακή διακυβέρνηση. Από το 2005 μέχρι το 2014, 1% των ε, Λιβανέζων, των πιο πλούσιων, έχουν το 1 τέταρτο του εθνικού πλούτου. Και στην ίδια περίοδο το 10% των πιο πλούσιων αύξησαν τα εισοδήματά τους 5 με 15%, ενώ οι πιο φτωχοί έχασαν το 1 τέταρτο των δικών τους εσόδων. Τώρα μεταξύ άλλων παραγόντων μπορούμε να αναφέρουμε επίσης και τη μεγάλη δημογραφική πίεση. Οι νέοι στο Λίβανο είναι το 41%, είναι κάτω δηλαδή από 24 ετών και πολλοί από αυτούς τους νέους είναι άνεργοι. Επίσης, τα προβλήματα αυτά της, που είναι δηλαδή χαμηλή η, η οικονομία της χώρας με την κακή διακυβέρνηση οδηγούν, όπως καταλαβαίνετε, σε μια κατάσταση διαφυγής εγκεφάλων. Φεύγουν οι νέοι από τη χώρα. Το δημοσιονομικό σύστημα επίσης έχει φτάσει στα ωριά του με τριπλό έλλειμμα. Δημοσιονομικό, 3 δισεκατομμύρια το 2018, δημόσιο χρέος, περίφημο 150% του ΕΠ, το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο και Έχουμε και δείκτες στο κόκκινο όταν μιλάμε για τις εμπορικές, το εμπορικό ισοζύγιο με 17 δισεκατομμύρια έλλειμμα το 18 και αρνητικό ισοζύγιο πληρωμών επίσης μείον 6,4 δισεκατομμύρια ε, δολάρια για τους πρώτους μήνες του 2019. Ποια είναι η συνέπεια ότι χάνει την εμπιστοσύνη του ο κόσμος και Βέβαια, πιέζεται και το νόμισμα και δημιουργείται και μια μαύρη αγορά με, όσον αφορά την ε, ε, συναλλαγματική τιμή απέναντι στο δολάριο. Από το 2018 ε, λειτουργούμε συνενετικά με κυβέρνηση εθνικής ενότητας από το 2013 και εφαρμόζει, εφαρμόζουν όλες οι δυνάμεις που είναι στην κυβέρνηση, εφαρμόζουν διάφορα μέτρα συνενετικά, κάτι το οποίο έχει βέβαια πλέον εκτήματα, έχουν πρόσβαση στους δημόσιους πόρους, κάτι το οποίο οδηγεί σε ολιγαρχία τελικά και ευνοεί όσους βρίσκονται πολύ κοντά στην πολιτική αυτή τάξη. Με αποτέλεσμα ο υπόλοιπο πληθυσμό να φτωχαίνει. Το 2015 ξεκίνησαν κάποιες διαμαρτυρίες εξαιτία της κρίσης των αποβλήτων, των σκουπιδιών. Γιατί μαζεύτηκαν σκουπίδια στους δρόμους της ε, Βυρίτου, κυρίως στο ανατολικό τμήμα, και έτσι ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες ε, τότε ε, σε σχέση με την αντικατάσταση της εταιρεία που μάζευε τα σκουπίδια τότε. Και πολιτικά είχε σημασία αυτό, γιατί δημιουργήθηκε μια νέα πολιτική, ένα νέο πολιτικό κόμμα το 2016 στις δημοτικές εκλογές στη Βηρητό. Είχαμε μια εναλλακτική ομάδα η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στο χώρο. Το 2018 εμφανίστηκαν και άλλα ψηφοδέλτια εναλλακτικά που όμως ε, κανένα δεν κατάφερε να αλλάξει την ε, κοινοβουλευτική σκηνή με λίγους βουλευτές και ανεξάρτητη πολιτικά. Φτάνουμε λοιπόν στις διαμαρτυρίες του 2019 το πολιτικό σύστημα παρέμεινε δρανέ. Δεν έκανε τίποτα, γιατί δεν είναι εξοπλισμένο να αντιμετωπίσει αυτούς τους νέους παράγοντες που είναι οι άνθρωποι στο δρόμο, παντού στο Λίβανο. Έτσι, το πολιτικό σύστημα αγνοεί τις εκκλήσει που γίνονται από τον κόσμο για αξιοπρέπεια. Αγνοεί πλήρω και καταστέλει επιπλέον. Θα σα τα πει και ο συνάδελφο. Και ο λόγος των πολιτικών επίσης δείχνει αδράνεια και δεν κάνει τίποτα για να ικανοποιήσει θετήματα των διαμαρτυρώμενων. Υπάρχει λοιπόν μια φλόγα που έχει ανάψει και είναι κάτι που έλειπε εδώ και καιρό στο Λίβανο, που είναι η συμμετοχή του κόσμου, της κοινωνίας των πολιτών. Όπως επίσης και η κατάρριψη κάποιων ταμπού όσον αφορά τους πολιτικούς ηγέτες, του αρίμα όπως τους ονομάζουμε εδώ πέρα, που θεωρώντουσαν κάτι το ιερό μέχρι τώρα, ταμπού. Επίσης, κινητοποιούνται τώρα και οι γυναίκες. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε πριν. Τι ζητούν λοιπόν τώρα όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται. Το πρώτο το πετύχαμε, να παραιτηθεί κυβέρνηση. 29 Οκτωβρίου το πετύχαμε αυτό. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη βέβαια είναι η δημιουργία νέας κυβέρνησης, πρόορες εκλογές επίσης και καταπολέμηση, σοβαρά όμως, της διαφθοράς και ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Κάποιοι από αυτούς που διαμαρτύρονται ζητούν και αλλαγή του συστήματος, την ε, κατάργηση να πάψει πια αυτή η θρησκευτική κατανομή, να μην παρεμβαίνει δηλαδή ο θρησκευτικό παράγοντα στη διακυβέρνηση. Η κυβέρνηση, όπως είπαμε λοιπόν, ε, παρετήθηκε και η επόμενη κυβέρνηση δεν κατάφερε να κρατηθεί παρά μία εβδομάδα μόνο γιατί είχε στην ημερήσια διάταξή του, στους στόχους της δηλαδή, κάποια στοιχεία τα οποία ήταν εντελώς ασυμβίβαστα με τα αιτήματα των διαδηλωτών. Ποιο είναι το σενάριο λοιπόν τώρα που έχουμε μπροστά μας. Υπάρχει μια διελκυστίδα που συνεχίζεται στους δρόμους. Έχουμε μια αρτισκληρωτική βασικά πολιτική τάξη. Σήμερα το βράδυ θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Και όσον αφορά τώρα την Ευρώπη, φυσικά και θέλουμε στήριξη για να ε, παραμείνει σε σταθερότητα ο Λίβανος. Και για τους ε, στόχους και τα αιτήματά μας φυσικά με κύριο αίτημα αποχή από κάθε εκμετάλλευση των ε, αντιπαραθέσεων των γεωπολιτικών, Ιράν πρώτο και καλύτερο, που ενισχύει την κρίση στη χώρα. Έπειτα, προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ασφάλεια για τους διαδηλωτές. Επίσης, η Ευρώπη μπορεί εδώ να παίξει κάποιο ρόλο όπως έχει παίξει και παλιότερα, ε, στηρίζοντάς μας οικονομικά, τεχνικά, να προετοιμαστεί ο, στρατός για να μπορεί να πλαισιώσει τους διαδηλωτές και να διατηρηθεί η δημόσια τάξη χωρίς υπερβολική χρήση βίας. Τέλος, στήριξη στον εκδημοκρατισμό εκ των κάτω στο Λίβανο. Και αυτό είναι ένας ε, πολιτικός στόχος ε, για το Κοινοβούλιο. Εγώ θα μιλήσω αγγλικά, εάν μου επιτρέπετε, γιατί μιλάω καλύτερα αγγλικά από γαλλικά. Καταρχήν, όπως είπε και ο δόκτωρ, peux continuer. Alors, ah. juste deux petites minutes pour euh, changer. Απλώς δύο λεπτάκια για να αλλάξουμε το κανάλι της μετάφρασης, εφόσον θα μιλήσετε αγγλικά. Ένα λεπτό για την ρύθμιση. Problem. Pas problème. think that we can restart. Νομίζω ότι μπορούμε να ξαναρχίσουμε, αλλά στα αγγλικά τώρα. Yeah. Is it okay? Okay, we can we can do it in English now. Yeah, we will have the translation. Τώρα να περάσουμε στα αγγλικά. Καταρχάς είμαι ο Τζορτ Ράνι από την LSF, τον Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία ιδρύθηκε το 1996 και χαίρομαι που μπορώ να ενημερώσω την Επιτροπή σας, την έχω ήδη ενημερώσει μάλλον με email πρόσφατα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Λίβανο. Θα βλέπετε ότι αυτό που συμβαίνει σε σχέση με τις διαμαρτυρίες και τις εκτάσεις που έχουν πάρει την έκταση που έχουν πάρει, δεν είναι κάτι που μας εκπλήσει. Παρόλο που ήταν απρόβλεπτο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ετών είχαμε σημειώσει σειρά από παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης, που εξηγούν τις διαμαρτυρίες των τελευταίων 26 ημερών. Ήταν μια κινητοποίηση που χρειαζόταν από καιρό. Δεν θέλω εδώ να πάρω θέση ούτε υπέρ ούτε κατά των διαμαρτυριών και των διαδηλώσεων, αλλά είναι σαφές ότι από την σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στο πέρασμα των ετών δεν έχει γίνει καμιά σοβαρή προσπάθεια για να προστατευτούν τα δικαιώματα των πολιτών. Κυρίως ήθελα να μιλήσω για την ε, διαμαρτυρία την ίδια για το δικαίωμα του ε, Εδώ ξεκινήσαμε από το Σεπτέμβριο με την αύξηση κατά 6 δολάρια στη μετάδοση δεδομένων του WhatsApp, την εφαρμογή και την αύξηση των τελών. Ξεκινήσαμε από τις 17 και 18 Οκτωβρίου με τις πρώτες διαμαρτυρίες και με πολλές βίες περιπτώσεις καταστολής και μάλιστα και βιαιότητες ε, κατά της δημόσιας περιουσίας και της τάξης. Το πρωί και την, το βράδυ της 18ης Οκτωβρίου είδαμε δύο σύρους οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σε ένα εργοτάξιο διότι κοντά έπιασε πυρκαγιά και δεν μπορούσαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το κτίριο οπότε έχασαν τη ζωή τους από τις αναθυμιάσεις. Επίσης υπήρξε δυσανάλογη χρήση βίας σε αρκετές περιπτώσεις. Ως ΕΝΙΦ θέλουμε να τηρηθεί το δικαίωμα του διαμαρτύρεστε και του διαδηλώνει και θέλουμε να ε, κοιτάξουμε τις 26 μέρες αυτές των διαμαρτυριών τι γίνεται. Υπάρχει αύξηση στην, ε, στο κατά πόσον έχουν γίνει δημοφιλείς οι διαμαρτυρίες, έχουν ξεπεράσει τα όρια της φυρητού και όπου υπάρχει οδικό δίκτυο έχουν ε, αρχίσει να βγαίνουν στο δρόμο διαδηλωτές. Ήταν πραγματικά μια έκπληξη να βλέπουμε ότι οι διαδηλωτέ δεν συγκεντρώνονται απλώ στη Βηρητό, στι ε, συνηθισμένε πλατείες όπου γίνονται διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες, αλλά σε σημεία που συνήθως δεν υπήρχαν τέτοιε κινήσεις. Σε πολλά προάστια και πόλεις υπάρχει κίνηση των πολιτών και είναι συμβολική σημασία ότι ο μεγάλο αριθμό ανθρώπων που βγει στους δρόμους Μιλάμε για τις περιοχές βόρεια της Βεριτού, που είναι συνήθως ήσυχε περιοχές. Είναι περιοχές όπου δεν υπάρχουν δράσεις και κινήσεις διαδηλωτών. Όμως οι αναλυτές και οι πολιτικοί επιστήμονες λένε ότι είναι μάλιστα περιοχές όπου οι πελατειακές σχέσεις ε, ευημερούν και δεν έχουν την τάση οι άνθρωποι να διαμαρτύρονται εκεί. Βλέπουμε όμως να υπάρχει έντονη διαμαρτυρία και αν αναλύσουμε τις τάσεις των διαδηλώσεων, οι περισσότερες αμφισβητούν την άρχουσα τάξη στο Λίβανο και θέλουν να συζητηθούν, θέλουν να τεθούν θέματα διαφθοράς, κακής ε, διακυβέρνησης, νεποτισμού και σε μεγάλο βαθμό οι αντιδράσεις των επίσημων θεσμών σε πολλές αυτές, από αυτές τις διαδηλώσεις και τις διεκδικήσεις ήταν ε, βίες. Διότι ακριβώς αμφισβητείται η νομιμοποίηση των κυβερνώντων και της άρχουσας τάξης. Γι' αυτό αντιδρούν έτσι βία. Τις τελευταίες 26 μέρες, σε μεγάλο βαθμό, βλέπουμε ότι οι διαδηλώσεις έχουν μετατοπιστεί ε, από γραμμική, αν θέλουμε να τα δούμε γραμμικά, χρονικά δηλαδή, Αρχικά ξεκινήσαμε με ειρηνική ε, διαμαρτυρία, αλλά αν δούμε τα γεγονότα μέρα με τη μέρα, βλέπουμε και ε, ακραία βία να έχει εκδηλωθεί. Ιδίως τη μέρα της παρέτησης του Πρωθυπουργού Χαρίρη και μια-δυο μέρες πριν Είχαμε και αντιδιαδηλωτέ που είχαν βγει στους δρόμους και ξυλοκόπησαν άλλους διαμαρτυρήτέ του κινήματος ουσιαστικά παραβιάζοντας το δικαίωμα της ειρηνικής διαδήλωσης και το δικαίωμα της ε, σωματικής ασφάλειας των ανθρώπων αυτών. Συσπηρώθηκαν και αναγκάστηκαν να πάνε σε άλλη πλατεία ε, οι άνθρωποι τους ακολούθησαν και τους ξυλοκόπησαν και εκεί, πράγμα που το γνώριζαν οι διοκτικέ αρχές και έκαναν τα στραβά μάτια. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι θεσμοί ε, της χώρας δεν καταφέρνουν να προστατεύσουν το δικαίωμα της ειρηνικής διαδήλωσης και διευκολύνουν την εκδήλωση αυτών των δύο φαινομένων. Ήθελα επίσης να πω για το θέμα του νόμου Γενικής Αμνηστίας που συζητήθηκε σήμερα στο Κοινοβούλιο και κατά πάσα πιθανότητα θα περάσει, τελικά αναβλήθηκε η ψηφοφορία στην επόμενη εβδομάδα. Εμάς μας ανησυχεί πολύ αυτός ο νόμος της Γενικής ε, Ασυλίας, γιατί είναι εδώ και έξι μήνες που γίνεται αυτή η προσπάθεια για να προσπαθήσουν να περάσουν αυτόν τον νόμο σε όλες τις συζητήσεις. Ε, στο Κοινοβούλιο. Αυτός ο νόμος, αυτό το νομοσχέδιο ε, αλλάζει τα δεδομένα της, ε, του κράτους δικαίου στη χώρα, ενισχύει την αίσθηση της ατιμορρησίας, του δικαιώματο να είναι κανεί ατιμόρυτο και προστατεύει το status quo. ουσιαστικά παρεμποδίζεται η δικαστική αρχή της χώρας από τις δράσεις των πολιτικών, τους Βουλής και του ε, Κοινοβουλίου, της άρχουσας τάξης. Αυτό επηρεάζει βεβαίως και εμάς και δεν μπορούμε να κάνουμε κανονικά τη δουλειά μας. 20.000 ε, εντάλματα σύλληψης, παράδειγμα αυτό, για εμπορία ε, αυτή τη στιγμή για διακίνηση ναρκωτικών αυτή τη στιγμή πρόκειται να ακυρωθούν με τον ε, νόμο αυτό. Τι ε, μέλλον λοιπόν μπορούμε να σχεδιάσουμε εάν δεν υπάρχει δυνατότητα για πολιτικές διαπραγματεύσεις Εάν μπορεί κανεί με παζάρια και ε, με πολιτικά παιχνίδια να πάρει κάποιο είδου αμνηστία, κάποιο είδου ασυλία και να αποφύγει το δικαστικό σύστημα, να το παρακάμψει τελείω. Και στα τελευταία λίγα λεπτά που έχω για το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω υπό το φω ε, του Συμβουλίου ε, και το τι μπορεί να γίνει σε σχέση με τις πρωτοβουλίες σας θα πρέπει να μην υπάρχει τόση επικέντρωση, τόση έμφαση στην αιρεσιμότητα και να κοιτάξουμε τι δυνατότητες επενδύσεις μπορούσαν να υπάρξουν. Οι πρόσφατες αλλαγές στο Λίβανο και υπό το φως των πρόσφατων δυναμικών που διαμορφώνονται μέσα από τις διαδηλώσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να στηρίξει να στηρίξει τους κατάλληλους φορείς, αλλά να δείξει και τη δέουσα επιμέλεια για το πώς θα έπρεπε να εκφραστεί ε, να λάβει σάρκα και οστά η αλληλεγγύη αυτή προς το, η υποστήριξη προς το Λίβανο για να, όχι για να ενισχυθεί ε, η άρξα τάξη και το status quo αλλά να λειτουργήσει εύρυθμα το σύστημα. Θα πρέπει να απαιτηθούν περισσότερες σοβαρότερες δεσμεύσει από το κράτος του Λιβάνου για το κράτο δικαίου, για τη λειτουργία της δικαστικής, του δικαστικού συστήματος και βάσει μιας μελέτης που έγινε πρόσφατα από το Λιβανέζικο Κέντρο για Πολιτικές Μελέτες Χρειάζεται δικαστική αρχή ανεξάρτητη για να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα που είδαμε πρόσφατα. Θα πρέπει στην κοινωνία των πολιτών να υπάρξουν περισσότεροι νόμοι που να προστατεύουν τους πολίτες και να εγγυώνται την ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής. Και παρόλο που εμ, πολλοί ήταν αυτοί που υποστήριξαν ένα τέτοιο νομοσχέδιο, τελικά δεν έφτασε ποτέ να προχωρήσει αρκετά στη Βουλή μας γιατί παρακολύθηκε και πήρε πάρα πολύ χρόνο. Χρονοτριβήσαν στο να την εξετάσουν την πρόταση. Thank Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να δώσω το λόγο τώρα στους βουλευτές. Δεν ξέρω ποιος θέλει το λόγο. Ο κύριος Γκέτα. Ένα ερώτημα θέλω να σας θέσω. Κάτι τη δικιά σας άποψη, ποια είναι τα ενδεχόμενα τις επόμενες 10-20 μέρες. Ραφαήλ Λούξμαν. Λούξμαν. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερος για την παρουσία σας στην εικονική εδώ και για το κουράγιο σας, το θάρρος σας μάλλον. Α, ήθελα να μου εξηγήσετε περισσότερο για το πώς θεωρείτε ότι το κίνημα αυτό δεν θα ε, ενταχθεί σε μια λογική που να προωθεί συγκεκριμένα θρησκευτικά συμφέροντα. Με ποιον τρόπο, μπορεί, με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο αυτό να καπελωθεί, αν θέλετε, από τις θρησκευτικέ αντιπαλότητες. Θα ήθελε κάποιο άλλο το λόγο, ρωτάει η Πρόεδρος, και αν όχι θα ήθελα να σας θέσω εγώ κάποιες ερωτήσεις. Για αυτό που είπατε, ότι πλέον έχουμε φτάσει στο τέλος ενός συστήματος που ε, βασιζόταν στην ισορροπία μεταξύ των θρησκευτικών ομάδων στο Λίβανο. Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, ποιο, τι μέλη ποιο είναι το επόμενο εναλλακτικό σύστημα και πώς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό με ποιες μεταρρυθμίσεις και αν είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις που ζητάει ο δρόμος, ε, οι διαμαρτυρόμενοι. Δεύτερον, δεν μιλήσατε για το ρόλο της αστυνομίας όσον αφορά την διατήρηση της τάξης στο Λίβανο. Είναι διαφορετική η συμπεριφορά, είναι διαφορετικά τα πρωτόκολλα εμπλοκής που χρησιμοποιούν σε σχέση με τη διατήρηξη της τάξης και σε σχέση με την στάση τους απέναντι στους διαδηλωτές. Το τρίτο μου ερώτημα έχει παρόμοιο με αυτό που σας έθεσε ο κ. Γκετά. Ποιες είναι οι προοπτικές για το μέλλον αναφέρατε ότι θα οργανωθούν ε, πρόορες εκλογές. Ποιες βλέπετε όμως να είναι προοπτικές του Λιβάνου μεσοπρόθεσμα. Δεν μιλήσατε και τόσο για το ζήτημα της μετανάστευσης, αν και αναφερθήκατε στην οικονομική κατάσταση όμω, αυτή τη στιγμή ε, είναι πολύ μεγάλο ο αριθμό των εκτοπισμένων των προσφύγων από τη Συρία, αλλά επίση και ο αριθμό των προσφύγων από την Παλαιστίνη που βρίσκονται στο Λίβανο. Θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι ο αντίκτυπο τη παρουσία των προσφύγων στη σημερινή κατάσταση στη χώρα σα. Τέλο, αναφερθήκατε στι ε, μεταρρυθμίσεις στην ε, Συμφωνία σύνδεση και το πόσο θα πρέπει να ξαναδούμε κατά πόσον μπορεί αυτή η Συμφωνία Σύνδεσης να συνεισφέρει στην εμπέδωση του κράτους δικαίου στο Λίβανο. Μήπως μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένοι και να μας δώσετε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις ε, από τη δική σας πλευρά για το πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε την ε, Συμφωνία ε, Σύνδεσης με την Ένωση. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τα μέλη του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής σας. ξεκινώ με την πρώτη τελευταία ερώτηση που μου θέσατε, δηλαδή για το ζήτημα της μετανάστευσης θα μιλήσω και το ζήτημα των προσφύγων από την Παλαιστίνη και τη Συρία που βρίσκονται στο Λίβανο. Πράγματι, ο στιγματισμός, η δαιμονοποίηση αυτών των ομάδων του πληθυσμού που πολύ συστηματικά ε, την διέπραξαν οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια και πολλές άλλες πολιτικές ομάδες. Οδήγησε στο να κατηγορούν τους πρόσφυγες για την κατάσταση με τους οικισμούς, την κατάσταση με τις υποδομές και πράγματι το γνωρίζετε ήδη, ο Λίβανος είναι η χώρα που έχει το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων σε σχέση με τον πληθυσμό του. Εδώ θα έλεγα ότι καταδεικνύεται πόσο πολιτικά όρημοι είναι εκείνοι που διαδηλώνουν. Γιατί δεν υπήρξε μια τέτοια σύγκρουση, δεν διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή ε, να απειλούνται ούτε άμεσα ούτε έμεσα οι πρόσφυγες. Δεν υπήρξε δηλαδή κάποια κίνηση εναντίον τους, έχουν μείνει ε, προστατευμένοι στην άκρη ξεχωριστά από όλη αυτή την σύγκρουση που ξεκίνησε με τις διαδηλώσεις. Δεν λοιπόν ε, ε, ευωδόθηκε αυτή η προσπάθεια να παρουσιαστεί ότι οι πρόσφυγες φταίνε για τα δεινά του Λιβάνου. Γνωρίζετε τον, τον αριθμό των ε, προσφύγων. Διαπιστώνουμε ότι τα τελευταία δέκα χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των Παλαιστινίων προσφύγων σχεδόν 220.000 120 ε, να βρίσκονται στη χώρα και να αντιμετωπίζουν μια σειρά προβλημάτων ανάμεσα σε αυτά διοικητικά προβλήματα, προβλήματα δηλαδή στη σχέση τους με τη δημόσια διοίκηση και προβλήματα ανεργίας. Γι' αυτό είναι μια ευχαριστή έκπληξη να διαπιστώνει κανεί ότι δεν του χρησιμοποιούν ω από δύο Πομπέου τράγου ούτε του Παλαιστίνιου πρόσφυγε ούτε του ε, Σύριου πρόσφυγε. Τώρα σε σχέση με την αστυνομία έχετε δίκιο, μίλησα πολύ περισσότερο για το στρατό. Βεβαίω, αποτελεί το αντικείμενο τη αστυνομία η διαχείριση των διαδηλώσεων και η διτήρηση τη ε, τάξη ιδιαίτερα όταν αυτές οι διαμαρτυρίες λαμβάνουν χώρο στο δημόσιο χώρο. Έχουν εξοπλισμό στη διάθεσή τους και δυστυχώς, όπως ο συνάδελφός μου κ. Ραλή το, σας το ανέφερε ήδη, διαπιστώνουμε τεράστια αύξηση της παράνομης βίας. Κάτι που έχουν ήδη καταγγείλει οι τοπικοί ακτιβιστές και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ταυτόχρονα βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι οι μονάδες του στρατού δεν είναι προετοιμασμένες για να αντιμετωπίζουν διαδηλωτές, δεν έχουν την αντίστοιχη ε, εκπαίδευση γιατί δεν είναι αυτός και ο στόχος τους εξάλλου. Και χρειάστηκε να προσαρμοστεί η εκπαίδευσή τους έτσι ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τους συναδέλφους τους στην αστυνομία. Και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό, αυτή η αποστολή στον στρατό του Λιβάνου έχει δοθεί από το 2010. Χωρίς βέβαια να, να τηρηθεί αυτό που τότε είχε λεχθεί ότι θα ήταν ένα προσωρινό μέτρο. Φαίνεται ότι αυτή η αλλαγή του χαρακτήρα του στρατού είχε μόνιμο, είναι μόνιμο, είναι μόνιμο χαρακτήρα. Έχει και κάποια άλλα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά αυτό το κίνημα διαμαρτυρίας. Πέρα από την κατάρριψη ορισμένων ταμπού, στην οποία ήδη αναφέρθηκα, αλλά είναι επίσης και το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε γέφυρες και να ξεπεράσουμε ε, ομαδοποιήσεις και χάσματα που υπήρχαν ανάμεσα στις διαφορετικές θρησκευτικέ ομάδες ή πολιτικές ομάδες ή κοινωνικές ομάδες. Παραδοσιακά στο Λίβανο αυτό χρησιμοποιείται το φόβητρο της θρησκευτική σύγκρουσης. Και οδηγούμαστε σε καταστάσεις όπου οι πολίτες περισσότερο να εμπιστεύονται εκείνον που ήταν ο θρησκευτικός του ηγέτης παρά τους συμπολίτε τους με τους οποίους ε, ε, περνούν τα ίδια δεινά σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Ε, λοιπόν, στο δρόμο αυτού, αυτές οι διαφορές γεφυρώθηκαν Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι η πλειοψηφία των Σουνιτών καταφέρνει να συνεννοείται με άλλες περιοχές, διαδηλωτές σε άλλες περιοχές που μπορεί να είναι κατά πλειοψηφία χριστιανοί. σιγά σιγά δηλαδή δημιουργείται ε, μια αίσθηση ε, ε, αλληλεγγύης η οποία βέβαια δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει να θεωρήσουμε ότι έχουν πάψει να έχουν σημασία οι υπόλοιπε ταυτότητε των πολιτών, η θρησκευτική του ταυτότητα, για παράδειγμα. Αλλά αναγνωρίζουν οι πολίτε του Λιβάνου όλο και περισσότερο ότι η θρησκευτική του ταυτότητα δεν είναι ασύμβατη με την ιδιότητά του ω πολίτε. Και ότι εν τέλει υπάρχουν κοινά συμφέροντα και ανάμεσα σε αυτά τα κοινά συμφέροντα είναι και η αρμονική συνύπαρξη των διαφόρων θρησκευτικών ομάδων. Εξάλλου, ο Λίβανος είναι ε, η χώρα η οποία κατεξοχήν έχει καταφέρει αυτή την συνύπαρξη των διαφόρων θρησκειών. Και το, την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων θρησκευτικών ομάδων. Προσπάθ, έγινε μια προσπάθεια αυτό να χρησιμοποιηθεί και στην ε, ε, στον καταπερισμό των διαφόρων εξουσιών στο πολιτικό σύστημα αυτή όμως απέτυχε. Ακριβώς αυτό είναι που προσπαθούμε τώρα να μεταρρυθμίσουμε. Και δυστυχώς μετά την αποτυχία αυτής της ε, κατανομής των εξουσιών οδηγηθήκαμε σε, αυξημένη, σε όλο και πιο αυξημένη διαφθορά που βλάπτει τα συμφέροντα όλων των πολιτών ανεξαρτήτως θρησκείας. Είναι δύσκολο λοιπόν να κάνει προβλέψεις κανείς σήμερα για το τι πρόκειται να συμβεί. αλλά διαβάζουμε στο Σύνταγμα του Λιβάνου το, από το 1800, ε, 1989 που έθεσε τέλος την εμφύλια σύγκρουση ε, στη Συμφωνία του Ταχέρ αναφέρεται ρητά τροπολογίες μάλλον του συντάγματος που πέρασαν το 1991, προ, προβλέπεται λοιπόν ρητά ότι θα υπάρξει μια μετάβαση από το σύστημα στο οποίο η πολιτική εξουσία κατανέμεται ανάλογα με τις θρησκευτικέ ομάδες. Θα περάσουμε σε μια εθνοσυνέλευση. Αυτή τη στιγμή γνωρίζετε ότι σήμερα υπάρχουν ποσοστώσεις, έτσι ώστε να υπάρχει ισότιμη εκπροσώπηση των χριστιανών και των μουσουλμάνων. Το άρθρο 22 όμως του συντάγματος προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση αυτού του συστήματος, η οποία εν τέλει θα οδηγήσει στη δημιουργία γερουσίας, που θα το αντικαταστήσει. Αν το δει λοιπόν κανείς από συνταγματικής απόψεως, ο δικός χάρτης είναι ξεκάθαρος. Το τι θα πρέπει να γίνει. Το ερώτημα βέβαια είναι εάν οι διάφορες πολιτικές ομάδες θα έχουν το πολιτικό θάρρος που χρειάζεται για να προχωρήσουν αυτή τη μεταρρύθμιση που θεωρώ ότι είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τη θρησκευτική ταυτότητα που είναι και αυτή ένα αναγνωρισμένο ανθρώπινο δικαίωμα από τη μια και την ε, δυνατότητα συμμετοχής στα κοινά που επίσης είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα που προστατεύεται και από το Σύνταγμά μας. Πολλοί από τους διαδηλωτές εξάλλου ζητούν να τηρηθεί η συνταγματική τάξη, Άλλοι είναι πιο ριζοσπάστες και πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα και ζητούν να καταργηθεί πλήρω ο καταμερισμό των πολιτικών αξιωμάτων με βάση το θρησκεύμα. Προβλέπω ότι το πιο πιθανό δυστυχώς θα είναι να συνεχίσουμε. Όπως σήμερα να έχουμε μια πολιτική ελίτ η οποία να, μην, να, να κοφεύει απέναντι σε όλες αυτές τις ε, απαιτήσει των διαδηλωτών. Φοβάμαι ότι θα υπάρξει όλο και μεγαλύτερη ριζοσπαστικοποίηση του κινήματος εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης και με λίγα λόγια, όσο περισσότερο περνάει ο καιρό, τόσο μεγαλύτερα είναι ο κίνδυνο να υπάρξουν εντάσεις και να οδηγηθούμε σε συγκρούσεις που να θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και την ασφάλεια της χώρας. Αυτό είναι το άσχημο σενάριο. Και αυτό λοιπόν πολλοί από τους διαδηλωτές απαιτούν από την, τους πολιτικούς ηθήνοντες να επιταχύνουν τις μεταρρυθμίσεις ακριβώς έτσι ώστε να λιγοστέψει αυτή η ένταση και να μπορέσει η ε, κοινωνία του Λιβάνου να επανέλθει στο δρόμο της, του εκδημοκρατισμού της χώρας. Επιτρέψτε μου να προσθέσω κι εγώ μερικά πράγματα. You Νομίζω ότι μπορείτε να συνεχίσετε. Καλώς. Έλεγα λοιπόν ότι από τη δικιά μου την πλευρά συμφωνώ σε πολλά με τον κύριο Μούφτη, αλλά έχω και κάποιες διαφορετικές απόψεις. Κυρίως από, επειδή από διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις ακούω ότι σε ένα βαθμό, κοιτάξτε εμείς προσπαθούμε να διαχωρίσουμε τα πράγματα δεν, ξέρουμε, δεν λέμε ότι θα υπάρξουν οικονομικές συνέπειες αν καταρρεύσει το πολιτικό σύστημα ή το οικονομικό. Δεν λέμε ότι θα υπάρξει περισσότερη διαφθορά και ευνοιοκρατία. Πάντως, η πολιτική ταυτότητας που έχουμε, που βασίζεται σε αυτό το θρησκευτικό κατά κάποιο τρόπο σύστημα θρησκευτικών κοινοτήτων, είναι ένας παράγοντας, αλλά δεν είναι ο μόνος. Και δεν θα ήθελα φυσικά να δημιουργήσω προσδοκίες ότι αν αλλάξει το σύστημα τότε θα λυθούν και όλα τα προβλήματα του Λιβάνου. Πολύ αμφιβάλλω, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Και άλλες χώρες στον κόσμο έχουν περάσει από κάτι τέτοιο. Έχουν τεράστια διαφθορά χωρίς ε, το θέμα της ταυτότητας. Ο Λίβανος πάντως έτσι κι αλλιώς έχει την υποχρέωση. Πρέπει να διορθώσει την κατάσταση, να προβεί σε μεταρρυθμίσεις, είτε αλλάξει το σύστημα είτε δεν αλλάξει. Δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο και η δικαστική εξουσία δεν έχουν την υποχρέωση να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις. Και επιτρέψτε μου να απαντήσω και στην πρώτη ερώτηση για τις πρώτες 10-20 μέρες. Πολλοί από τους φίλους μου και από τους συναδέρφους επί 26 μέρες με επικρίνουν ότι είμαι πάρα πολύ ρεαλιστής και συνεχίζω νομίζω και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνω για να με εντάξει και απέναντί σας. Έτσι λοιπόν τώρα πιστεύω ότι αυτό που γίνεται δεν είναι ότι υπάρχει κάποια αντιμετώπιση της κρίσης, υπάρχει παρέτηση του Χαρίρη θυμόσαστε ότι είχαν γίνει εκλογέ το 2016 και στη συνέχεια κατέρευσε η κυβέρνηση. Τώρα γίνονται διαπραγματεύσεις για ένα νέο πρωθυπουργό, αλλά είναι διαπραγματεύσεις για μια νέα εξουσία. Οι μεταρρυθμίσεις, η καταπολέμηση της διαφθοράς και της ευνιοκρατίας είναι κάτι το οποίο φυσικά και χρειάζεται αυτή η αλλαγή αλλά τα πολιτικά κόμματα δεν συζητούν για μεταρρυθμίσεις, δεν διαπραγματεύονται ε, για δαπάνες, αλλά για μια νέα συμφωνία εξουσίας. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό. Οπότε πρέπει να δούμε μετά τις 17 Οκτωβρίου τι βλέπουμε. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο στο Λίβανο ήταν ειρήνη, ασφάλεια το 2015 σε μικρότερο βέβαια βαθμό είδαμε το περιβάλλον και αντιμετώπιση της ρήπανση. Τώρα έχουμε το θέμα της διαφθοράς και της ευνοιοκρατίας που κυριαρχεί στο σκηνικό. Πάντως για τις επόμενες 10-20 μέρες που ρωτάτε τι περιμένουμε. Με την αποτυχία των διαπραγματεύσεων του Νοεμβρίου του 2016 τι έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Δεν πρόκειται μόνο για μεταρρυθμίσεις, πρόκειται για τις εκλογές που θα έχουμε το 2022, για τις ε, συμμαχίες που θα συμμετέχουν στις εκλογές αυτές. Έχουμε επίσης και προεδρικές εκλογές το 2022. Οπότε τι θα γίνει, θα έχουμε ένα νέο κενό, γιατί με τόσο σημαντικά ζητήματα ε, μεταρρυθμίσεις, προεδρικές εκλογές, ε, κοινοβουλευτικές κτλ. Είναι πολλά πράγματα προς συζήτηση. Και αν συζητηθούν υποποίηση, δεν ξέρω κατά πόσο θα παραμείνει η σημερινή κατάσταση ή όχι. Τώρα τι μπορεί να κάνει Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της Συμφωνίας Σύνδεσης. Ένα σημαντικό είναι να επανακαθορίσει την ιερεσιμότητα. Δηλαδή, εκείνοι οι οποίοι δικαιούνται στήριξη και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αμφισβητούνται βέβαια όπως και από την κοινωνία και το κοινοβούλιο αλλά το ίδιο θα πρέπει να γίνει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην δηλαδή υπονομευθεί το σύστημα ελέγχων ε, του Λίβανου αλλά να βεβαιωθούμε ότι λειτουργεί. Είναι μια χώρα που τα τελευταία 30 χρόνια οι έλεγχοι αυτοί δεν πήγαν καλά, οπότε βασιζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι και δωρητής μας να παίξει το ρόλο της. Ω κοινωνία των πολιτών πιέζουμε και το δικό μας κοινοβούλιο και τη δικαστική μας εξουσία να παίξουν αυτό το ελεκτικό ρόλο. Αλλά αυτό που πρέπει ακόμα να γίνει είναι να υπάρξει και αλλαγή στην θεωρητική σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Λίβανο. Δυστυχώς η θεωρία της αλλαγής βασίζεται σε σταθερότητα. Δηλαδή αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, στήριξη των υπηρεσιών ασφάλειας, ε, το μεταναστευτικό. Δυστυχώς όμως δεν βλέπουμε αυτή την θεωρία να βοηθάει το Λίβανο. Αν βάζετε υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και προϋποθέσεις, τότε καταλήγουμε σε μια αρνητική, θα έλεγα εγώ, σταθερότητα. Έτσι την ονομάζω εγώ. Και όχι μακροπρόθεσμα σταθερότητα. Και επειδή υπάρχει και το θέμα του νόμου για την αμνηστία. Όταν δεν είναι ανεξάρτητο το δικαστικό σώμα, όταν υπάρχουν πρακτικέ βασανισμών, ε, καταχρηστικέ ε, κρατήσει, ε, κακέ συνθήκε στι φυλακέ, οι οικογένειε των φυλακισμένων διαμαρτύρονται εδώ και τρία χρόνια και ζητάνε να απελευθερωθούν οι αγαπημένοι του. Η λύση της κυβέρνησης δεν είναι να διορθώσει τη δικαστική εξουσία, όχι να κρατήσει ε, αυτούς που φταίνε, δεν είναι να σταματήσει καταχρηστικές ε, και κτλ, αλλά αμνηστία. Και το μοντέλο σταθερότητας δεν είναι ε, πρότυπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα η δικιά σας επιτροπή θα μπορούσε να επανακαθορίσει τη σχέση αυτή με το Λίβανο, με πρακτικές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να φροντίσει η σταθερότητα που χρειάζεται ο Λίβανος δεν έχει να κάνει με τις υπηρεσίες ασφάλειας ή τους αξιωματούχους, αλλά με την βελτίωση της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από το 2015 έχουμε δει πάνω από αυτά ανθρώπου να έχουν πεθάνει από βασανισμού, χωρί να υπάρχει λογοδοσία. Τα τελευταία 7 χρόνια επίση υιοθετήθηκε ένα νόμο σχετικά με του βασανισμού, αλλά τελικά δεν πήγε καμία υπόθεση στη δικαιοσύνη για να καταδεκαστούν οι βασανιστές. Επίσης υπάρχει και ένας νόμος για ένα όργανο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά η κυβέρνηση δεν θέλει να το χρηματοδοτήσει. Πριν από μερικούς μήνες κανείς δεν είχε αναλάβει. Οπότε όλα αυτά θέτουν ερωτήματα. Πόσο στα σοβαρά παίρνει τα ανθρώπινα δικαιώματα τελικά ο Λίβανος. Και αυτό πρέπει να ε, συμπεριληφθεί στις προτεραιότητες. Ενώ στις προτεραιότητες του 2016-2020 βλέπετε ότι υπάρχουν οι στόχοι και οι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ε, μικρότερε από αυτέ που βάζει ο Λίβανος. Αυτό θα πρέπει να αντιστραφεί δεδομένη τη κατάσταση στο Λίβανο. Πρέπει να δεσμευτεί ο λίβανο ότι θα κάνει περισσότερα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δείκτε πρέπει να ξεκαθαριστούν περισσότερο τι δηλαδή αναμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το Λίβανο και ο Λίβανος πρέπει να παρουσιάζεται περισσότερη διαφάνεια Ποιο είναι το ποσοστό της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, τι κάνει ο Λίβανος για να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση. Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση στους πολίτες δεν το λέω αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για την κυβέρνηση του Λιβάνου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γκετά θέλει να ξαναπάρει το λόγο. Ναι, εάν μπορώ να σχολιάσω τις απαντήσεις σας. Ούτε ως υπενιγμό, ούτε μεταξύ των λεγόμενων σας δεν αναφέρατε κάτι το απεσιόδοξο. Η χρήση βίας από τους πολιτικούς και στρατιωτικούς του Λιβανέζικου συστήματος δεν φαίνεται να κινείται από ξένες δυνάμεις εμέσως ή απευθείας. Δεν θέλετε να φανείτε απεσιόδοξοι και γι' αυτό δεν λέτε κάτι τέτοιο. Ή θέλετε να παραμένετε στα πλαίσια όσων θεωρούνται αρμόζοντα και πρέποντα. Διότι οι ισορροπίες δυνάμεων σήμερα στο Λίβανο δεν αποκλείουν ίσως βραχυπρόθεσμα, μάλλον φαίνεται να αποκλείουν βραχυπρόθεσμα μια τέτοια εξέλιξη. Έχετε το λόγο. Να ξεκινήσω απαντώντας απλώς το εξή. Δεν είναι να αποκλείεται κάποιο απεσιόδοξο σενάριο. Και εγώ και ο κύριος Μούφτη μιλήσαμε για την αβεβαιότητα της τελευταίες ημέρες όταν οι Λιβανέζοι μιλάνε για αβεβαιότητα το θεωρούν και αυτό πηγές οπισοδοξία. Αλλά εμείς είδαμε τη βία στους δρόμους Είδαμε το τι συμβαίνει. Είδαμε ότι κάποιοι διαδηλωτές βγαίνουν στους δρόμους για να ξυλοκοπήσουν άλλους. Τους λένε ότι δεν επιτρέπεται να διαμαρτύρονται και την ίδια μέρα βλέπουμε να γίνονται όλα αυτά με την ανοχή των ε, δικτικών αρχών, της αστυνομίας. Αυτό είναι ένα έμεσο μήνυμα ότι η βία επιτρέπεται η αστυνομία ε, υποτίθεται ότι σας προστατεύει, αλλά άμα θέλει μπορεί και να σταματήσει να σας προστατεύει. Αλλά υπάρχει και ο νόμος περί αμνηστίας, περί ασυλίας. είναι ένα απτό αποδεικτικό στοιχείο, πιστεύω. Η αμνηστία, ακόμα και σήμερα, εάν γινόταν κανονικά η Σύνοδος στη Βουλή, ε, υπήρχαν διαδηλωτέ στου δρόμου που είχαν βγει για να του εμποδίσουν ακριβώ να πάνε ω εκεί και να ψηφίσουν για τον νόμο αυτό. Οι πολιτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν του μπλοκαρισμένου δρόμου για να στείλουν στου υποστηρικτέ του το εξή μήνυμα. Εμεί θέλουμε να βγάλουμε τα παιδιά σα από τη φυλακή, να του δώσουμε ασυλία και αμνηστία. Θέλουμε να ε, ακυρώσουμε και να αναστείλουμε τα εντάλματα σύλληψη που ισχύουν για 10.000 ε, ανθρώπου, αλλά δεν μα αφήνουν οι διαδηλωτέ που έχουν κλείσει του δρόμου. Τι μήνυμα είναι αυτό, ε, ότι υπάρχουν κάποιοι αρχηγοί σε φυλές, σε φρατρίες που μπορούν να ωφεληθούν από το νόμο αυτό περί ασυλίας και να ε, απηχήσουν το μήνυμα αυτό στους διαδηλωτές τους δρόμους για να φτάσει αυτό και ως απόϊχο στη Βουλή. Το λέω για το επίπεδο πόλωσης που παρατηρούμε αυτή τη στιγμή στις διαδηλώσεις στους δρόμους. Και αυτό μας ανησυχεί. Το να περάσει αυτή τη στιγμή ο νόμος περί αμνηστίας με όλους τους διχασμούς και τις ε, που υπάρχουν στο λιπανέζικο λαό ε, θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και στην Τρίπολη οι άνθρωποι που έχουν πάρει μέρος στις διαμαρτυρίες τελευταίες 26 μέρες πραγματικά μπορεί να οδηγήσει στο να μην τα βρίσκουν μεταξύ τους οι γιατί κάποιον τα παιδιά είναι ακόμα στη φυλακή. Δεν ξέρω αν ο κύριος Μουφτή έχει διαφορετική άποψη για το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Όντως, το απεσιόδοξο σενάριο όλοι το σκέφτονται, αλλά γιατί δεν το αναφέρουμε ρητός. Δεν το κάνουμε για να μην ε, γίνει από προκατάληψη, αλλά από την άποψη της εξουσίας, αν κάναμε μια πολιτολογική ανάλυση και από διεθνής άποψη του τι συμβαίνει, αυτό που συμβαίνει είναι και η συμβαστική λύση που βρέθηκε για το προεδρικό αξίωμα το 2016. Και Το σύστημα αυτό κατανομής των εξουσιών ε, οδήγησε και στην ανάληψη εξουσιών του κυρίου Αρών στο ε, ύψιστο αξίωμα. Ήταν ένας πολιτικός συμβασμός αυτός. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, ο Πρωθυπουργός που προσπάθησε να χειραγωγήσει τους διαδηλωτές, να τους εκμεταλλευτεί ξεκάθαρα, παρατήθηκε. Και αφήνει την ευθύνη στους πολιτικούς του αντιπάλους. Εάν μιλήσουμε λοιπόν για το σενάριο που αναφέρατε και εσείς, εγώ θα το απέφευγα αυτό, δεν θα το έπαιρνα ως πρώτη επιλογή. Είναι λίγο δύσκολο να αποδώσουμε συγκεκριμένε προθέσει σε όσου δρούν αυτή τη στιγμή ε, διότι φαίνεται να επιδιώκουν την ανανέωση του προεδρικής αυτής συμβαστική λύση, ε, εφόσον τουλάχιστον ε, οι διαδηλωτέ τους δρόμου δεν έχουν καταφέρει να βρουν διαβλό ώστε να ακουστεί και σε πολιτικό επίπεδο η φωνή τους. δηλαδή ουσιαστικά αγνοούν πλήρως αυτά που λένε οι διαδηλωτές στους δρόμους είναι άλλη πολιτική μέρημνα. Ο καθένα θέλει να διαπραγματευτεί με βάση τα συμφέροντα των περιφερειακών υποστηρικτών του, των ε, αρχηγών σε φιλωτικό επίπεδο και να παραμείνει το status quo. Όμω εδώ το status quo φαίνεται να είναι αδύνατο, είναι ψεύδο ψεύδο καθεστώς ψευδοκαθεστική ατάξη, γιατί η διαμαρτυρία στους δρόμους δεν τα αφήσει αυτό να γίνει. η τοποθέτηση του Λιβάνου σε σχέση με το Ιράν ε, έχει ρίξει όλο το βάρος το ότι θα υπάρξει κόπωση στις ε, διαμαρτυρίες και στο επίπεδο των διαδηλωτών. Οπότε δεν θα χρειαστούν σοβαρές μεταρρυθμίσεις, αλλά περισσότερο λαϊκιστικές ε, ως προς την μεταρρύθμιση και την ανα διοργάνωση του δικαστικού συστήματος, το φορολικό και ούτω καθεξής. Διότι η πολιτική τάξη ουσιαστικά εξηγεί τα όσα συμβαίνουν ως τώρα. Το 2005 μέχρι το 2005 μάλλον η Συρία ουσιαστικά επηρέαζε τα πράγματα, τις πολιτικές υποθέσεις στο Λίβανο. Από το 2005 στο 2011 η Συρία και η Σαουδική Αραβία επηρέαζαν επίσης τα πράγματα χάρη στους ε, πολιτικούς τους συνεργάτες σε περιφερειακό επίπεδο στην, ε, στο Λίβανο και από το 2011 έχει βγει από το προσκήνιο η Συρία και έχει πατήσει πόδι το Ιράν. Οπότε από το 2012 βρισκόμαστε απευθείας αντιμέτωποι με την αντιπαράθεση Ιράν με τη Δύση και ένα ρόλο ολένα αυξανόμενα ε, της Σαουδικής Αραβίας που ξέρετε ότι ουσιαστικά εκβίασε τον ε, Λιβανέζο Πρωθυπουργό ε, το 2017 διότι ήταν ακριβώς ε, αγανακτισμένη με τις παραχωρήσεις που έκανε ο Λιβανέζος Πρωθυπουργός στο Ιράν. Με αυτές λοιπόν τις εξελίξεις και αν τα ξαναδούμε από το φως των σημερινών εξελίξεων, όλοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα γεγονότα στους δρόμους, τις διαμαρτυρίες, για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους τα ίδια πολιτικά συμφέροντα με τον χαρακτήρα αυτόν, τον ε, τοπικιστικό και τον ε, θρησκευτικό που έχουν. βέβαια, είδαμε ότι ενώ έχει παρατηθεί ο Πρωθυπουργό δεν υπάρχουν ε, διαπραγματεύσει σε επίπεδο Βουλή. Γιατί? Γιατί ακριβώς ε, γίνονται αλλιώς οι συνεννοήσεις. Αυτό λοιπόν που θα μπορούσα να σας απαντήσω είναι ότι η σειροπία των δυνάμεων οδηγεί στο να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μην χαθούν τα πάντα. Δεν νομίζω όμως ότι έχουμε φτάσει ακόμη στην άκρη του γκρεμού. Ναι, και απλώς να συμπληρώσω όπως οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανησυχούν για το πώς θα βρεθεί μια νέα συμβαστική λύση και αναρωτιούνται ποια θα είναι η αντίδραση των πολιτικών εθνοντών, πώς θα κινητοποιήσουν τις ε, διεκτικές αρχές και πώς θα υλοποιήσουν αυτή τη νέα συμβαστική λύση. Αυτό που πραγματικά μας ανησυχεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το τι θα συμβεί με το δικαίωμα του διαδηλώνει. Η συμβαστική λύση κατά πάσα πιθανότητα θα σημαίνει ότι θα επιβληθεί κάτι σε όλους. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ για τι ε, τις παρουσιάσεις σας, κύριε Μουφτή και κύριε Χαλή. Ε, θα παραμένουμε σε επιφυλακή για να παρακολουθούμε το τι συμβαίνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Λίβανο. Ευχαριστούμε πολύ για τη παρουσία σα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και τώρα ο λόγο στην, Επιτροπή Εξωτερική, στην Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για να κλείσουμε τη συζήτηση. Uh, Ξωτήμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέλω να σας ευχαριστήσω ε, πρόσκληση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένου μα για την πολύ ειλικρινή και πλήρη καταγραφή και περιγραφή της κατάστασης στο Λίβανο. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Ήδη αναφέρθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εδώ και 40 χρόνια μια πολύ ισχυρή σχέση με το Λίβανο, η οποία έχει εκφραστεί με τη Συμφωνία Σύνδεση και τι σχετικέ προτεραιότητε. Υπάρχει και η αντίστοιχη χρηματοδότηση, η οποία ανέρχεται σε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2011, δηλαδή από την αρχή τη κρίση στη Συρία. Αναφερθήκατε επίσης στις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης και οι οποίες πράγματι τονίζουν την σημασία που έχει να ενισχυθεί η λειτουργία της δημοκρατίας και η χρηστή διακυβέρνηση. Έχουμε, μια συνεχή, ε, έχουμε ένα συνεχή διάλογο με τις λιβανικές αρχές για τα ζητήματα της διακυβέρνησης. Έχουμε επίσης και προγράμματα ε, βοήθειας, παροχής βοήθειας τεχνικής προς την κυβέρνηση αυτή, έτσι ώστε να τηρηθούν αυτές οι υποχρεώσεις. Μετά από τις πρόσφατες διαδηλώσεις, διαπιστώνουμε ότι πάλι αυτό γίνεται επ' ευκαιρία μιας ε, ανησυχητικής οικονομικής κατάστασης και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει ότι η υλοποίηση των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που να φέρουν κοινωνική δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Ζητούμε επίσης να γίνεται διάλογος χωρίς αποκλεισμούς για να εφαρμόζονται αυτές οι μεταρρυθμίσεις και αυτό που κάνουμε τώρα είναι μέρος αυτού του διαλόγου. Τονίζω λοιπόν και πάλι ότι αναγνωρίζουμε πόσο απογοητευμένο είναι ο λαό του Λιβάνου που ζητάει λογοδοσία και που ζητάει η κυβέρνησή του να ανταποκριθεί σωστότερα στι ανάγκε του. Με αυτήν τη λογική και με αυτό το σκεπτικό θα προσεγγίσουμε μια νέα κυβέρνηση που ευελπιστούμε ότι θα αναδειχθεί έτσι ώστε να μπορέσει αυτή να υλοποιήσει τι σχετικέ μεταρρυθμίσει. Βλέπω δεν έχω και πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, επομένω θα περιοριστώ σε αυτά. Σα ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Πρέπει να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ε, σας αποχαιρετούμε τους δύο προσκύκλημένους από το Λίβανο. Γεια σας. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, όπως έλεγα, ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθείται αυτή τη στιγμή για ζητήματα επιχειρήσεων και ανθρωπινών δικαιωμάτων και την 7η ε, Σύνοδο της Ανοιχτής Διακυβερνητικής Ομάδας Εργασίας για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, το 8ο ε, ετήσιο φόρουμ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καλωσορίζουμε την κυρία Ντενίζο Κλέαχ, η οποία είναι σύμβουλος της οργάνωσης ΣΥΝΤΣΕ, μια οργάνωση η οποία συμμετείχε στις διάφορες συζητήσεις που έγιναν στη Γενέβη και η οποία θα μας παρουσιάσει την οπτική γωνία της μη κυβερνητική οργάνωσης που εκπροσωπεί για αυτές τις εξελίξεις, για αυτό το διάλογο στην Γενέβη. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο Μπέρντ Λάγκ και τον κύριο Τόμπε από τις Επιτροπές Ίντα και Ντέβε αντιστοίχω, με τους οποίους είχα τη χαρά να, ε, με τους οποίους έχω τη χαρά να συμπροεδρεύω σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. Βεβαίως πρόκειται για ένα ζήτημα που είναι προτεραιότητα για την ε, Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι ένα θέμα επίσης πολύ σημαντικό για, σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε νομοθεσία στη Γαλλία, για παράδειγμα στην Ολλανδία για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας, για την καταπολέμηση του τράφικινγκ. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν αναλευθεί στη Βρετανία ή επίσης και στη Γερμανία. Και επίσης η φινλανδική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να περάσει υποχρεωτική νομοθεσία για την δέουσα επιμέλεια που πρέπει να επιδεικνύουν οι επιχειρήσει σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Λοιπόν, γίνονται αλλαγέ και γίνονται πρόοδοι, σημειώνονται πρόοδοι στον τομέα αυτό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να συζητήσουμε τι συζητήθηκε σε αυτήν την ε, πέμπτη σύνοδο της ανοιχτή διακυβερνητική Ομάδα για τις διεθνικές επιχειρήσεις και άλλες επιχειρήσεις σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα που διοργανώθηκε τον Οκτώβριο του 2019 συζητήθηκε το ενδεχόμενο να αναθεωρηθεί η συνθήκη η οποία συμφωνήθηκε τον Ιούλιο του 2019. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμετείχε στις αυτές τις διαπραγματεύσεις, μιας και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν, έδωσε, δεν στην Επιτροπή την αντίστοιχη εντολή διαπραγματεύση. Ωστόσο, η συμφωνία αυτή είναι πλήρως συμβατή με τις αρχές που έχει υιοθετήσει ο Οργανισμός ε, Ηνωμένων Εθνών για το ρόλο των επιχειρήσεων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγώ προσωπικά εκπροσωπώντας το ε, συμμετείχαμε στις διαπραγματεύσεις για την δημιουργία αυτής της νομικά δεσμευτικής συνθήκης και τονίσαμε την σημασία που έχει η πιο ενεργό συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρώπη, των Περιφερειακών Κοινοβουλίων στην Ευρώπη, καθώς επίσης και των Κοινοβουλίων της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής. Όλα αυτά εντάσσονται σε μια παγκόσμια εκστρατεία για να σταματήσει η ατιμορρυσία, για να ενισχυθούν τα δικαιώματα και η εθνική κυριαρχία των πολιτών έναντι αυτών των, διεθνών, ε, των πολυεθνικών επιχειρήσεων εκπροσωπήθηκαν ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές, τοπικά κοινοβούλια, πάνω από 100 ε, βουλευτές και συζητήθηκε το θέμα λοιπόν της δημιουργίας μιας νομικά δεσμευτικής συνθήκης για το ζήτημα. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Λάγκ, ο οποίος έχει ήδη ασχοληθεί με το ζήτημα της δέουσας επιμέλειας στο πλαίσιο των Συμφωνιών Διεθνούς Εμπορίου και μετά στο συνάδελφο από την Επιτροπή Ντέβε για να μας μιλήσει για τις σχέσεις του ζητήματος με την ανάπτυξη. Κύριε Λάγκε. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Με ιδιαίτερη χαρά μου δίνεται ευκαιρία να συζητήσω μαζί από κοινού με την Τρουά και την Τέβε για αυτό το θέμα. Εμείς πάντα ζητάμε δέους επιμέλεια, πάντα θέλουμε ισότιμη κατάσταση και πάντα θέλουμε να υπάρχουν σαφείς προοπτικές για την καταπολέμηση των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και είναι γεγονός ότι η εθελοντική βάση δεν έχει οδηγήσει σε αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε για τη δέουσα επιμέλεια σε αυτήν ε, την ε, αλυσίδα ε, προμήθειας σε όλα τα στάδια και κυρίως Υπάρχουν εθελοντικά προγράμματα για το χρυσό για παράδειγμα, αλλά ένα πολύ μικρό ποσοστό από το ρηκτά καλύπτεται. Γι' αυτό λοιπόν ζητήσαμε δέος επιμέλεια από τις επιχειρήσεις, από την εξόριξη μέχρι την πώληση χρυσού. Μέχρι που φτάνει στα δαχτυλίδια σας. Έτσι λοιπόν να καλύψουμε όλη την αλυσίδα των ορυκτών και θέλουμε αυτή τη δέουσα επιμέλεια σε όλη την πορεία. Έτσι λοιπόν, ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις το 2014 στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών για να υπάρξει μια δεσμευτική συμφωνία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κλάδο. Δυστυχώς δεν υπάρχει εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Πολλές φορές το έχουμε ζητήσει. Και οι χώρες μέλη πάντα είχαν κάποιον ε, υπουργό που ζητάει εντολή ώστε να είμαστε ενεργά μέλη και όχι απλώς παρατηρητές. Δυστυχώς όμως δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μετά από την τελευταία μας συνάντηση πριν από ένα χρόνο, αν δεν απατώμε. Έγιναν τον Οκτώβριο συζητήσεις και πολύ θα ήθελα να γνωρίζω τα αποτελέσματα. Και ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί περισσότερο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή αυτή. Ένα δεσμευτικό μέσο το οποίο θα μπορούσε να ρυθμίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στις δραστηριότητε διεθνούς συνεργασίας είναι ένα ζήτημα που απασχολεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και πολλά χρόνια ήδη. Από το 2014 όταν είχαμε την εντολή του ε, Συμβουλίου στον ΟΗΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, παρακολουθεί τις εξελίξεις, τις διαπραγματεύσεις και τις συμμετοχές. Από το 2014 και μετά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει την διακυβερνητική διαδικασία που κατέληξε σε νέα διαφορετικά κοινοβουλευτικά ψηφίσματα με το τελευταίο του Οκτωβρίου του 2018 όπου αναφέρεται η δυνατότητα μιας δεσμευτικής συμφωνίας από τον ΟΙΕ. Τώρα είμαστε στην πέμπτη σύνοδο τη Διακυβερνητική Ομάδα Εργασία για τι εθνικέ Εταιρείε και άλλε επιχειρήσει και ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε περιμένουμε τα αποτελέσματα. Και θέλουμε να ακούσουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, όλο ιδιαίτερο, για ό,τι εξελίξει υπάρχουν προ αυτή την κατεύθυνση μια δεσμευτική συμφωνία. Γνωρίζουμε επίσης ότι κάποιες χώρες μέλη έχουν εκφράσει ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται διαπραγματεύσεις μέχρι τώρα. Οπότε θέλουμε ενημέρωση και να δούμε κατά πόσο έχουν αντιμετωπιστεί αυτά τα ζητήματα μέχρι σήμερα ή όχι. Επίσης θα ήθελα πολύ να ακούσω και τις δικές σας σκέψεις για το πώς βλέπετε εσείς να προχωράει αυτή η διαδικασία από εδώ και πέρα. Θα συμμετέχει το Κοινοβούλιο σε μια νέα εντολή Περιμένουμε λοιπόν περισσότερα. Ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο κατευθείαν στην Τενής, η οποία θα μας ενημερώσει για τις μη κυβερνικές οργανώσεις. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τη δυνατότητα αυτή που μου δίνετε. Πρώτα απ' όλα, η συζήτηση αυτή έχει να κάνει και με το πρώτο ε, σημείο στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής αυτής χτες, όταν είχατε ανταλλαγή απόψεων με τις ε, γυναίκες που ε, δουλεύουν για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι γυναίκες αυτές ε, φυσικά και θα πρέπει να προσεχθούν περισσότερο γιατί ασχολούνται με τις ευθύνες των εταιριών ακριβώς. Η ΣΥΤΣΕ είναι μια οργάνωση ομπρέλα για μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Από το 2005 ε, λειτουργούμε και έχουμε διάφορες συμφωνίες και ασχοληθήκαμε και με τις ρυθμίσεις όσον αφορά την εξόριξη ορυκτών και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως επίσης τη δέωση επιμέλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σίγουρα υπάρχουν πιέσεις, σίγουρα δικαιώματα παραβιάζονται, ε, σίγουρα όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τη γη και με τα τρόφιμα. Τώρα όταν κάποιος δουλεύει για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θέλει να βοηθήσει για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να πάει επί τόπου και εκεί βλέπει ότι υπάρχει μια διελκυστίδα ε, εξουσιών και ε, δύναμης. Όλα αυτά συνδέονται περιβάλλον, ανθρώπινα δικαιώματα, κλίμα, γη, εργασιακά δικαιώματα, επενδύσεις, ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Και στις δικές μας οργανώσεις έχουμε βοήθεια και από το 2015 ε, με βοήθεια από γιατρούς, ε, από ανθρώπους που δουλεύουν για τον Αμαζόνιο και βλέπουμε τελικά ποιες είναι οι τάσει. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι υπάρχουν βασικές αρχές που, στις οποίες βασίζεται η δικιά μας η δράση και δεν ε, είμαστε υπέρ του ή του άλλου. Ε, κοιτάμε όλες τις πλευρές, την ε, επιμερισμένη ευθύνη, γιατί είναι πράγματα τα οποία μας αφορούν όλους. Επίσης, την υπεύθυνη εργασία για υπεύθυνε επιχειρήσεις που λογοδοτούν. Και επίσης θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι οικονομικοί παράγοντες και τα οικονομικά συμφέροντα μάλλον δεν είναι υπεράνω του ανθρώπινου παράγοντα. Έχουμε λοιπόν δουλέψει για μια εμβληματική περίπτωση που ήταν κάτι που καταδείξαμε και στη Σύνοδο της Γενέβης και αυτό είναι οι καταστροφές που έλαβαν χώρα στην Βραζιλία το 2015 και το 2019 που καταστράφηκαν φράγματα στο Μαριάννα και στο Μπουριντίνιο. Και μας επισκέφθηκαν και ακτιβιστές από τις περιοχές αυτές. Το 2015 ήταν μια από τις χρονιές της χειρότερης καταστροφής περιβαλλοντικής για τη Βραζιλία και το 2019 επανελήφθηκε και υπάρχουν και άλλα φράγματα που βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Είναι μόνο στη Βραζιλία αυτά? Όχι. Πρώτα είχαμε ένα άλλο στο οποίο συμμετείχε και η BHB μαζί με μια βραζιλιάνικη εταιρεία και είναι η πρώτη δικαστική περίπτωση στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί συμμετείχε και αυτή η Αυστραλιανή εταιρεία. Και μετά στο Πρεμεντίνιο ήταν μια γερμανική εταιρεία, η οποία έχει επιβεβαιώσει ότι είναι ασφαλές το φράγμα αυτό πριν καταρρεύσει. Και κάποιες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επίσης είχαν χρηματοδοτήσει εξορυκτικές δραστηριότητες, είχαν αγοράσει ε, το σίδερο ή άλλα υλικά τα οποία είχαν εξορυχθεί εκεί. Οπότε πρέπει να υπάρχει ο χώρος στο βήμα για να συζητηθούν αυτά. Δεν είναι μόνο για τη Βραζιλία, τα ξέρετε και στη Γαλλία. Είχαμε την έκρηξη στη Ρουάν ε, τα τους τελευταίους μήνες. Πρόκειται για μια αμερικανική επιχείρηση, η Λουμπριζόν, το εργαστήριο εκεί, κάτι το οποίο πλήττει ολόκληρη την περιοχή της Ρουάν. Νομικά ποιος είναι υπεύθυνο όμως και ποιος θα αποζημιώσει για την κατάσταση. Οπότε με αυτό, αυτό το πλαίσιο πρέπει μετά να στραφούμε και στο τι γίνεται ε, στα πλαίσια της ε, συμφωνίας του ΟΗΕ και ποιες είναι οι προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Γενέβη είδαμε ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή της διαδικασίας. Για πολλά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγε ότι η διαδικασία δεν είναι βιώσιμη και δεν συμμετείχε. Βλέπαμε βέβαια ότι συμμετείχε σε άλλα διεθνή φόρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πρόοδο της αναθεώρησης των δικαιωμάτων των επενδυτών, για παράδειγμα, και των διεθνών μηχανισμών ε, που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των επενδυτών. Και τον Οκτώβριο είναι ενδιαφέρον. Συγχρόνω γινόντουσαν διαπραγματεύσει ε, στη Γενέβη και στην ε, Βιέννη και για το εμπορικό δίκαιο και για το περιβάλλον για τους μηχανισμούς δηλαδή αυτούς ε, για τους επενδυτές και βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στην αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε αυτά τα δύο. Δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο πολυμερές ε, πλαίσιο με ό,τι γνωρίζουμε ενώ με τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει αποσυρθεί η Αμερική, η ομάδα εργασία είναι μια ομάδα εργασία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν πολύ καλό να συμμετέχει και εκεί. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέροντε καιροί για την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν δύο διαφορέ στο σχέδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει προ την κατεύθυνση αυτού που ζητάει και το αναφέραμε. Έχει να κάνει με την συνέπεια απέναντι στι αρχέ του ΟΗΕ. Και το άλλο έχει να κάνει με το πεδίο εφαρμογή του μέσου, που δεν θα καλύπτει μόνο διασυνοριακέ ε, δραστηριότητε, αλλά και στο εσωτερικό των χωρών. Θα τα καλύπτει όλα δηλαδή. Συνεπώς υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη όσον αφορά τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν αφισβητεί πια αυτή τη διαδικασία και μάλιστα εξέφρασε ικανοποίηση απέναντι στον Πρόεδρο και αναγνωρίζει ότι έχει, έχουν γίνει βήματα προς τα μπρος ώστε να έχουμε μία προσέγγιση που να μπορεί να υποστηριχτεί από πολλέ χώρε μέλη. Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε κάποιε διευκρινήσει. Και κάτι άλλο ενδιαφέρον είναι ότι πολλέ χώρε μέλη παρενέβησαν στη διαδικασία αυτή. Η Ισπανία, η Γαλλία και το Βέλγιο. Και αυτό αντικατοπτρίζει και το γεγονός ότι οι περιοχές που καλύπτονται από τη συνθήκη είναι επιμερισμένης αρμοδιότητας άλλες Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλες χωρών μελών. Και στην ε, τελευταία συνεδρίαση της Συνόδου είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε τη δυνατότητα της κοινωνίας των πολιτών να μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία, γιατί άλλες χώρες πίεσαν προκειμένου να μειωθεί ο χώρος στον οποίο μπορούν να παρέμβουν ε, εκπρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών και να μπορούν να παρεύουν μόνο οι χώρε μέλη. Αυτό που είναι ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι πολλά από τα θέματα που αποτελούν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αντικατοπτρίζονται στο ίδιο το μέσο, στι συζητήσει δηλαδή για το περιεχόμενο τη συνθήκη. Πρόσβαση σε αποζημίωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει, όπως και άλλοι, ότι εδώ υπάρχει μια δυναμία από πλευρά των Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η συνθήκη μπορεί να αποτελέσει προστιθέμενη αξία όσον αφορά εταιρείε και ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει στο αναθεωρημένο σχέδιο μια πρόταση για να υπάρχει νομική ευθύνη από τις χώρες. Και επίσης αναφέρονται και τα εμπόδια όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία και τις επαφές, θέμα ε, δικαιοδοσίας, τι μπορούν να κάνουν τα δικαστήρια δηλαδή. Συνεπώς, αυτό είναι ενδιαφέρον στοιχείο. Ένα άλλο ενδιαφέρον είναι η πρόληψη. Γίνονται συζητήσεις για τη δέωσα επιμέλεια που σίγουρα εμπνέονται από τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες μέλη και αποτελεί μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει τη συζήτηση αυτή σε διεθνές επίπεδο εκ παραλλήλου με τις συζητήσεις οι οποίες εξελίσσονται και λαμβάνουν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα, υποστηρικτέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό έχει να κάνει και με το πρώτο σημείο χτε στην ημερήσια διάταξη τη Επιτροπή σα. Το σχέδιο έχει διατυπώσεις οι οποίες αναγνωρίζουν ότι χρειάζονται μηχανισμοί για καλύτερη προστασία των υποστηρικτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των αυτόχθονων κοινοτήτων, για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, για αποτελεσματική συνένεση κλπ. Πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Και τέλος, υπάρχουν και συζητήσεις για το πώς το μέσο αυτό θα συνδέεται με συμφωνίε εμπορικέ και επενδυτικέ. Εκ παραλίλου λοιπόν προχωρούν αυτά τα ζητήματα, γι' αυτό είναι κάτι που σαφώς και ενδιαφέρει όλους ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, όσον αφορά τις παρατηρήσεις μας, να ξέρετε ότι γίνεται σοβαρή νομική συζήτηση για να δούμε τι μπορεί να προχωρήσει σε διεθνές επίπεδο και η συζήτηση γίνεται με πυρογνώμονες που λαμβάνουν υπόψη τους και τα εθνικά νομικά πλαίσια. Λαμβάνεται πίσει στο διεθνές πλαίσιο, διεθνεί δομέ. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν 90 χώρε οι οποίε συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση. Συνεπώ, κοιτάμε όχι μόνο τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχει και εδώ ένας χώρος ε, από τον οποίο μπορούμε να πιέσουμε πολλέ χώρε, τη Βραζιλία αλλά και πολλέ άλλε. Γιατί πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει περισσότερο στη διαδικασία. Όσο προχωράμε περισσότερο στι διαπραγματεύσει και τις συζητήσεις, μόνο οι χώρες που παρεμβαίνουν θα διαμορφώσουν τελικά το μέσο αυτό. Η Ρωσία και η Κίνα πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ καλά προετοιμασμένες. Και από πλευρά ε, των κοινοτήτων με τι οποίε δουλεύουμε, πραγματικά εκφράζουν μεγάλη απογοήτευση που δεν δραστηριοποιείται περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηρίξει ε, πράγματα τα οποία του ενδιαφέρουν και του αφορούν όπω η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα περιβαλλοντικά δικαιώματα, οι περιβαλλοντικέ αποζημιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Το δεύτερο είναι ότι αναφέρθηκαν ε, τα μέσα, τα νομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή εδώ είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο μπορεί να προσφέρει εμπειρία η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ξέρει από τέτοια νομικά μέσα και μπορεί να τα φέρει στα διεθνή φόρα. Και επειδή υπάρχουν προσδοκίες. Υπάρχει και κινητοποίηση πολλών φορέων. Πάνω από 270 ε, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών ήταν στην Γενέβη που αποτελούν μια συμμαχία και πιέζουν για να υλοποιηθεί μια τέτοια συνθήκη και πιέζουν και τα διεθνή συνδικάτα. Υπάρχουν επίσης και από την Εκκλησία εκπρόσωποι ακαδημαϊκοί που κινητοποιούνται κλπ. κλπ. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, όσον αφορά τις εταιρείε και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το σχετικό φόρουμ δηλαδή, υπάρχει συμπληρωματικότητα εδώ, ανάμεσα στις κατευθυντήριες γραμμές και τη συνθήκη. Βέβαια, προς το παρόν, δεν έχουμε προχωρήσει σε νομικά πλαίσια. Υπάρχει εδώ περιθώριο για συζήτηση και πρέπει να γεφυρωθούν τα δύο. Τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομίζω ότι πολλά έχει κάνει ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά σα. Ε, βλέπετε τα πράγματα από πλευρά διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Προσπαθείτε και εσεί να καθορίσετε τι προτεραιότητες τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα υπάρχει αντιπροσωπεία των Ευρωβουλευτών που συμμετείχε και είναι πολύ σημαντικό όλες αυτές οι πλευρές να συμμετέχουν. Κάποιες ε, πλευρές που θέλουν να συμμετέχουν τον Οκτώβριο δεν μπόρεσαν, αλλά νομίζω ότι στην επόμενη σύνοδο που προβλέπεται για το 2019 ελπίζω να μπορέσουν. Έπειτα η ΚΟΣΟΚ, η Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή, ετοιμάζει μία δήλωση, είχε ακρόαση για τέτοια θέματα. Οπότε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να φροντίσει να προωθήσει το έργο της ΕΚΟΣΟΚ, της ΟΚΕ δηλαδή. Έπειτα θα υπάρξουν και άλλα πράγματα που θα γίνουν. Νομική ανάλυση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει ήδη. Δεν ξέρω αν τα ξέρει αυτά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα σας ενδιαφέρει φαντάζομαι και στα επόμενα βήματα να υπάρξουν διαβουλεύσεις, υπάρχουν προθεσμίες για τη διαδικασία της συνθήκης, 30 Νοεμβρίου για τις τελικές παρατηρήσεις μετά από τον Οκτώβριο και παρατηρήσεις για το δεύτερο αναθεωρημένο σχέδιο. Στο μεταξύ υπάρχει και ο προπολογισμό που πρέπει να επιβεβαιωθεί. Ζωτική σημασία και αυτό το σημείο που θα έρθει το Δεκέμβριο. Και νομίζω τέλος ότι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να δει τι θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η νέα της ηγεσία θα πρέπει να βάλει αυτά τα θέματα στην ημερήσια της διάταξη. Έχουμε και ένα ε, ψήφισμα εδώ με συγκέντρωση υπογραφών να σταματήσει η εκστρατεία και ελπίζω να μπορέσουμε να σας παραδώσουμε ε, τα ψηφίσματα με τις υπογραφές ε, αυτές και σε εσά και στο Συμβούλιο. Και να ληφθεί υπόψη σε όλα τα επίπεδα και σε επίπεδο της συνθήκη, αλλά και σε επίπεδο της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε Ντενίζ, ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Και τώρα λόγος στους συναδέλφους που επιθυμούν να μιλήσουν. Η κυρία Χάουταλ έχει ζητήσει το λόγο. Mm. Ευχαριστώ εγώ ήθελα να ακούσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράχτη. Είναι εδώ, εφόσον είναι. Αλλά τέλο πάντων να πω ότι δεν υπάρχει θέμα. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε υποχρεωτική ιδέουσα επιμέλεια για τι ε, αλυσίδε τροφοδοσία. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι ευρωπαϊκέ εταιρείε δεν έχουν καμία συμμετοχή σε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραπεροντικέ ε, ζημιέ και φθορέ και ακούσαμε πολλά παραδείγματα στην Επιτροπή μας προσφάτως, όχι μόνο από τις σημερινέ παρουσιάσεις. Είναι λοιπόν ε, αυτονόητο αυτό. Και επίσης χαίρομαι που τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρεται να κινείται προς την κατεύθυνση όπου πιθανώς τα κράτη-μέλη θα αναθέσουν εντολή στην Ένωση ώστε να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσει τώρα κιόλας διεξοδική ανάλυση του σχεδίου που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο, αλλά ακόμα υπάρχουν αμφισημίε. διότι μιλήσαμε για νομική ευθύνη, πράγμα που σημαίνει ότι οι ορισμοί θα πρέπει να είναι πολύ αυστηροί, να μην παραμένει καμία ασάφεια για το τι είδου ε, επιπτώσει θα υπάρχουν από αυτέ του είδου τι ευθύνε. Θα ήθελα λοιπόν να μα πούν η ΕΕΔ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άποψή τους για το αναθεωρημένο σχέδιο πεδίου, το τι θα καλύπτει δηλαδή η συνθήκη. Και κυρίως για τα ανθρώπινα δικαιώματα. αυτό το σκέλος, η συνθήκη, τι εννοεί ακριβώς. Μιλά για όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά πώς πρέπει λίγο να διευκρινιστεί αυτό. Μήπως να μιλάει για όλα τα διεθνώς εγγυημένα προστατευόμενα ανθρώπινα δικαιώματα και ούτω καθεξής. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια σημεία που είναι λίγο ακατανόητα, όπως για την ευθύνη των εταιριών. Εάν δούμε τις σημερινές αλυσίδες τροφοδοσίες. Κάποιες είναι ιδιαίτερα περίπλοκες. Κάποια από τα πλημελήματα και τις ε, παρατυπίες κρύβονται ακριβώς σε διαφορετικούς κρίκους της αλυσίδας τροφοδοσίας. Θα πρέπει λοιπόν ίσως να υπάρχει κάποια είδους ανείχνευση της ευθύνης, ώστε και οι υπεργολάβοι και εκείνοι από πλευρά τους να μπορούν να αγγίθουν ότι δεν υπάρχουν παρατυπίες, παρανομίες ή οτιδήποτε παράτυπο. Και όχι μόνο να κοιτάζουμε την ευθύνη τη κυρίω υπεύθυνη εταιρεία. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα το πολύ σημαντικά στοιχεία αυτή τη συμφωνία να τα δούμε κατά λεπτό. Και επίση να πω εν τέλει ότι ακούσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσφέρει με τα δικά τη μέσα σε αυτές τις δημοτεύσει. ναι, αλλά διότι τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που μπορούμε να έχουμε ευρωπαϊκό εργαλείο για τη δέωση επιμέλεια. Δεν πρέπει να την χάσουμε αυτή την ευκαιρία, ούτε να αφήσουμε τι δύο αυτέ εξελίξει να λειτουργήσουν μία ει βάρο τη άλλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι πολύ ισχυρή στι διεθνεί διαπραγματεύσει, αλλά αν κάνουμε σωστά τη δουλειά μα στο εσωτερικό, μπορούμε να επιτρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, κοιτάξει τη σωστή εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών που έχουμε ήδη εγκρίνει όλοι εμεί και να ξεκινήσουμε από το δικό μα το επίπεδο. Ευχαριστούμε. Μιγγέλ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ περίμενα να ακούσω πρώτα τις τοποθετήσει τοποθετήσεις της Επιτροπής πριν να λάβω το λόγο, γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη ε, θέση της Επιτροπής και κυρίως τι πρόκειται να λάβει, ως να εκφράσει ως ε, θέση. Είναι καλό το, καλή είδηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραστεί στις ε, διαπραγματεύσεις, αλλά να δούμε αν αυτό τελικά είναι καλό ή κακό νέο, γιατί πρέπει να δούμε ποια θα είναι και η θέση που θα προωθήσουμε. Αυτή τη στιγμή η θέση που έχει ακουστεί να προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ταιριάζει με αυτή των κοινωνικών εργονώσεων. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτό που οι μη κυβερνητικέ οργανώσει προωθούν, αλλά επίση και αυτό που έχει ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λαμβάνει μια θέση η οποία να είναι συμβατή με τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό πολύ θα ήθελα να ξέρω τι σκοπεύει να λάβει ω θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι διαπραγματεύσει αυτέ. Γιατί φοβάμαι ότι θα πάμε ακόμα πιο κάτω από έναν κοινό παρονομαστή που είναι ήδη πολύ χαμηλό. Μιλούμε τώρα για ε, ζητήματα που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είχαν λυθεί στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Οργανισμού Εργασίας. Και χρησιμοποιούνται αυτά τα, αυτές τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα έπρεπε να μας πηγαίνουν πιο μπροστά, σε, ως εργαλείο εναντίον των διεκδικήσεων των δικών μας κοινοτήτων. Για παράδειγμα, μας θα πρέπει να φροντίσουμε να μην χρησιμοποιηθεί αυτή η συμφωνία τελικά προς όφελος των πολυεθνικών εταιριών και εναντίον εκείνων που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να μην χρησιμοποιηθεί τελικά αυτή η συμφωνία για να δικαιολογηθούν και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή είναι μια σημαντική ανησυχία που έχω, γι' αυτό θεωρώ πολύ σημαντικό να ακούσω τη θέση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστούμε πολύ, Μικέλ Ειρήνα. Ευχαριστώ. Απλώς να προσθέσω δύο πράγματα που είπε η κυρία Χάουταλα. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική δέσμευση στις ελληνικές τροφοδοσία, Αναφέρατε ότι μια σειρά από νομοθεσίες ευρωπαϊκών κρατών μελών θα πρέπει να κάνουν κάτι γι' αυτό, όπω το Ηνωμένο Βασίλειο πριν από λίγα χρόνια πέρασε το θέμα για την σύγχρονη δουλεία ε, στα εργασιακά. Και από τη δική μου προσωπική εμπειρία, στην προηγούμενο επαγγελματικό μου βίο εργάστηκα σε αυτό το τομέα και φαίνεται ότι έχουμε κάποια καλά αποτελέσματα από όσα έχουμε δει τουλάχιστον εμεί ω τώρα. Θα έπρεπε λοιπόν να το λάβουμε αυτό υπόψη, ιδίω ότι αφορά το τελευταίο κομμάτι της αλυσίδας τροφοδοσίας. Το άλλο θέμα είναι η εμπορία των ανθρώπων και η προσφορά, η παροχή υπηρεσιών, κάτι που μπορεί να συμπίπτει με την συγχρονή δουλεία και το σχετικό νόμο. Με ενδιαφέρει λοιπόν να μου πείτε αν υπάρχει κάτι γι' αυτό στο νέο σχέδιο συνθήκης. Ευχαριστώ, Νταν. Ναι, ε, για την ΕΕΔ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να μου πείτε εάν στη Ρωσία και την Κίνα είναι σωστές οι ανησυχίες για το σχέδιο τη συνθήκης, διότι δεν το αναγνώρισαν καν και δεν το δέχτηκαν ως βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Η δική σας η αποτίμηση ποια είναι, τι προβλέπετε να κάνουν. Και μετά, η πιο κοντινή μας εμπορική εταίροι, εάν μιλάμε για εμπόριο που βασίζεται σε εμπορικές ε, τιμές, ο Καναδάς και η Ιαπωνία δεν ήταν ούτε εκείνοι παρόντες. Υπάρχει κάποιος λόγος Ευχαριστώ. Έχω εγώ και δύο ερωτήσει. Πρώτα απ' όλα στην ΣΥΤΣΕ και μετά στην ΕΕΔ. Μιλάμε πολύ στο πολυμερές επίπεδο για την έλλειψη ισοτιμίας. Εμείς πάντοτε προασπιζόμασταν την πολυμερή προσέγγιση ως Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε για τη διεθνές εμπόριο, είτε για την COP21, δηλαδή για το περιβάλλον και το κλίμα. Εδώ βλέπουμε μια σχετική επιφυλακτικότητα για να πάμε προς το πολυμερές επίπεδο. Ε, πώς βλέπετε σε αυτές τις επιφυλάξεις, τους ενδιασμούς της Ευρώπης να, πάνε, να πάμε προς το προς την πολυμερή προσέγγιση και μετά για ένα ευρωπαϊκό εργαλείο, για μια ευρωπαϊκή διευθέτηση του θέματος της δέουσας επιμέλειας. Ε, θα μπορούσε αυτό να χρησιμοποιηθεί ως ένα συμπλήρωμα για το ε, παγκόσμιο εργαλείο, το διεθνές εργαλείο που θα μπορούσε να σχεδιαστεί για το θέμα αυτό και μετά για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Και εκεί βλέπουμε ότι σε επίπεδο 100 μελών υπάρχουν κάποιες κινήσεις. Τέσσερα με πέντε κράτη έχουν ήδη προ προτείνει κανόνες ε, και νομοθεσία για την ε, εταιρική ευθύνη εδώ. Όμως, σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως ε, η ΦΙΤΖΕ και οι εθνικοί φορεί. Είδαμε και συναντήσαμε εκπροσώπου εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του κακάο. Και θέλουν κανόνε, θέλουν νόμου. Διότι λένε ότι αν τώρα δεν υπάρξουν νόμοι, δεν υπάρξουν συγκεκριμένοι κανόνε, θα τα βρουν σκούρα. Εδώ λοιπόν η δημιουργικότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πώ μπορεί να αξιοποιηθεί. Συνήθω η Επιτροπή δεν περιμένει την εντολή του Συμβουλίου. Ε, σχεδιάζει, καταρτίζει νομοθεσία και την προτείνει, την υποβάλλει ω πρωτοβουλία στο Συμβούλιο. Για το θέμα λοιπόν αυτό το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, πώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει συντάξει ούτε μία μόνο μονοσέλιδη, θα έλεγα, πρόταση. Όπω έχει γίνει με την με το TTIP και τη σχετική εντολή. Εντάξει, συζητήσαμε μια από τι πιο σημαντικές εμπορικές συμφωνίες ε, ποτέ. Πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αξιοποίησε αυτήν την δυνατότητα εφευρετικότητας που έχει για να συντάξει έστω και ένα μονοσέλιδο έγγραφάκι προς το Συμβούλιο που να μπορέσει να ε, κάνει κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να στηρίξω τη δικιά σας την ερώτηση, γιατί και εγώ αναρωτιέμαι γιατί δεν υπάρχει εντολή όταν κοιτάω άλλες διεθνείς ε, εμπορικές διαπραγματεύσεις, συχνά, ε, πολύ γρήγορα είμαστε με εντολή. Οπότε εδώ πού είναι το πρόβλημα. Είναι κάποιες χώρες μέλη που δεν τη θέλουν και ποιες. Γιατί μια που έχουμε ήδη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι θέλουμε να δεσμευτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, ε, γιατί δεν έχουμε την εντολή. Είναι κάποιες χώρες που δεν θέλουν να συμμετάσχουμε ή κάτι άλλο είναι το πρόβλημα, για να ξέρω. Και στη συνάντηση που είχαμε στην Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου συζητήσαμε την εμπορική συμφωνία με το Βιετνάμ. Και θέλω να το πω και εδώ, ότι πραγματικά από τη μια μεριά προστατεύουμε τους, ε, τους επενδυτές, από την άλλη μεριά, όταν ερχόμαστε στα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν προχωράμε, ενώ για την προστασία των επενδυτών, ναι, προχωράμε. Υπάρχει μια ανισορροπία εδώ. Ωραία. Η ΣΥΤΣΕ πρώτα και μετά Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Δράση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη. Για το ερώτημα για το, γιατί υπήρξε διστακτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω επειδή στο το 2014 προτιμούσε να προωθήσει τις κατευθυντήριες αρχές της. Γι' αυτό το λόγο αυτή η διαδικασία ίσως να θεωρήθηκε ότι στόχευε ιδιαίτερα κάποιες πολύ μεγάλες πολυεθνικές αντί να έχει μια συνολική προσέγγιση. Όμως έτσι όπως έχει εξελιχθεί τώρα το νομικό μέσο, δεν πιστεύω ότι υπάρχει πια αυτό ο κίνδυνο ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Και θα έλεγα επίσης ότι το γεγονός ότι επί τέσσερα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκούσε κριτική σε αυτή τη διαδικασία οδήγησε σε κάποιε κάποιες χώρες να είναι και αυτές απρόθυμες να συμμετάσχουν. Αυτή τη στιγμή που έχει υπάρξει μια μεταστροφή λοιπόν της θέση τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευελπιστούμε ότι και οι χώρες αυτές θα είναι πιο πρόθυμες να συμμετάσχουν και επίσης χρειάζεται και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να απευθυνθεί προς τις χώρες αυτές και να τους ζητήσει να συμμετάσχουν καλόπιστα. Τώρα όσον αφορά τις... Στην οργάνωσή μας εργαζόμαστε και για τα δύο αυτά ζητήματα. Και θεωρούμε ότι και οι προσπάθειε της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, δέουσα επιμέλεια και η συμμετοχή της στις διαπραγματεύσεις για την ε, συνθήκη είναι απαραίτητες. Γιατί ήδη διαπιστώνουμε πρωτοβουλία σε εθνικό επίπεδο, στη Μεγάλη Βρετανία, στις κάτω χώρες. Όμως για μας το σημαντικό είναι αυτές οι διαδικασίες να τελεσφορήσουν και να ε, συνεχίσουν να προχωρούν συντονισμένα γιατί θεωρούμε ότι μπορούν να υπάρξουν συνέργειες. Δεν το είχα πει πιο πριν, αλλά πιστεύουμε ότι αυτές οι συζητήσεις που γίνονται ε, σε σχέση με την νομικά δεσμευτική συνθήκη οδηγούν και σε προόδους στο ευρωπαϊκό επίπεδο ή επίσης και στο εθνικό επίπεδο. Ε, βοηθούν δηλαδή και την ευρωπαϊκή νομοθεσία να βελτιωθεί, αλλά και, και σε άλλα επίπεδα η νομοθεσία να βελτιωθεί. Τώρα λοιπόν που ε, θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα να συμμετάσχει στη διαδικασία αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιστοίχω να ε, αρχίσει να εξετάζεται και η νομοθετική πρόταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον και την δέουσα επιμέλεια. Ο εκπρόσωπο τη ε, Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Συμφωνώ πλήρω με την κυρία Χάουτελα, με τον κύριο Λάγκε, που είπαν ότι η δέουσα επιμέλεια λειτουργεί ως Έννοια, έχω την τιμή να είμαι και πρόεδρος της ομάδας του ΟΑΣΕ για τα ματωμένα διαμάντια για τις, ε, τους πολύτιμους λίθους από εμπόλεμες περιοχές και βλέπω πως μπορεί να λειτουργήσει μια τέτοια διαδικασία στην οποία συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να δούμε όμως ποια θα είναι και τα επόμενα βήματα. Θα το έχετε πληροφορηθεί, θα το έχετε διαβάσει, ορισμένοι από σας βρίσκονταν και στην Γενέβη ότι κατά την εναρκτήρια δήλωσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επεσήμανε κάποιους κινδύνους. Κάποιους από αυτούς τους ανέφεραν ήδη η, κυρία, τους ανέφερε ήδη η κυρία Χάουτελα. Δηλαδή παραμένουν ανοιχτά ζητήματα σε αυτό το προσχέδιο συνθήκης και επίσης συνεχίζουμε να μην έχουμε διαπραγματευτική εντολή. Όμως θεωρούμε ότι το να καταλήξουμε σε ένα νομικά δεσμευτικό διεθνές κείμενο έχει προστιθέμενη αξία και μπορεί να συνεισφέρει στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξασφαλίζοντα επίση ότι αυτό θα γίνεται και χωρί τρέβλωση του ανταγωνισμού, όπω πολλοί από εσά ανέφεραν. Προσπαθούμε λοιπόν πολλέ από τι ανησυχίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να τι εισάγουμε σε αυτή τη συζήτηση, όπω για παράδειγμα την κάλυψη όλων των ε, νομικών προσώπων ή να φροντίσουμε η συνθήκη αυτή να είναι συμβατή με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και όλοι γνωρίζουμε ε, και το είπαν και κάποιοι από τους συμμετέχοντες στη Γενέβη, είναι πολύ δύσκολο κανείς να κάνει copy-paste σε ένα νομικό κείμενο από κατευθυντήριες αρχές σε νομικά δεσμευτικό κείμενο. Ε, σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι καταφέραμε να αφήσουμε πίσω μας και να ξεπεράσουμε τις ιδεολογικές διαφορές ή προσεγγίσεις. Συμφωνώ λοιπόν με την κυρία Οκλέχ ότι σε γενικές γραμμές οι παρεμβάσεις δεν είχαν συγκρουσιακό χαρακτήρα και προσωπικά χαίρομαι για το γεγονό ότι μπόρεσε να συμμετάσχει και να συνδεθεί το όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την τελική έκθεση αυτής της Συνόδου. Το ερώτημα βέβαια είναι, που θα πρέπει να μας αποσχολήσει, είναι ότι αυτή τη φορά έγινε για δεύτερη μόνο μόλις φορά μια πραγματική διαπραγμάτευση, ήρθαμε πιο κοντά σε ένα διεθνέ νομικό κείμενο το οποίο να έχει πραγματικά προστιθέμενη αξία, αλλά επίσης και να μπορεί να εφαρμοστεί και να επιβληθεί η εφαρμογή του. Το τρίτο, εξίσου σημαντικό και δύσκολο, να βρεθεί ένα νομικό κείμενο το οποίο να μπορεί να τύχει της υποστήριξης από χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, είτε αναπτυγμένες είτε αναπτυσσόμενες. Ε, και γι' αυτό θα υποβάλω στην Επιτροπή σας και στις τρεις Επιτροπές σας μάλλον, ότι Παρά το γεγονό ότι κατά τη διάρκεια τη Συνόδου ακούσαμε πολλέ παρατηρήσει, ε, διευκρινίστηκαν πολλά ζητήματα, θα υποβάλω την ιδέα ότι ακόμα παραμένει πολλή δουλειά να γίνει μέχρι να φτάσουμε στο επόμενο προσχέδιο, το οποίο προβλέπεται, όπως είπε και η κυρία Οκλέρ, τον Ιούνιο του 2020. Και ε, απομένει ακόμα πολλής δρόμος να καλυφθεί μέχρι να φτάσουμε σε ένα κείμενο το οποίο να μπορεί να αποτελέσει πραγματικά αντικείμενο διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων, τις πραγματικές δύσκολες διαπραγματεύσεις δηλαδή. Και όπως το φαντάζεστε δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα ο δρόμος για αυτές τις διαπραγματεύσεις. Το ανέφερε ήδη και ο κύριος Λάγκη. Ήδη όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της συνθήκης, η ομάδα των αφρικανικών κρατών επιμένει στη θέση της να καλύπτονται μόνο οι πολυεθνικές εταιρείες. Η Κίνα τοποθετήσε με την ίδια θέση σε σχέση με το άρθρο 5 και γενικά δεν θέλουν να προβλεφθεί, προβλεφθεί οποιαδήποτε υποχρέωση ως επιμέλειας όταν το, τη σύμβαση την έχει συνάψει η κυβέρνηση. Δηλαδή να φροντίσουμε οι αρχές αυτές να αφορούν μόνο τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Καντιλαμβανόμαστε γιατί το κάνει αυτό η Κίνα. Αλλά βλέπετε ότι έχει μια δύσκολη στάση. Ε, γιατί η Ρωσία είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιληφθεί κανείς αν πραγματικά επιθυμεί να εμπλακεί σε επί της ουσίας συζήτηση. και φοβάμαι ότι ανεξαρτήτως από το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπω να αλλάξει η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και φοβάμαι ότι σε μια παρόμοια κατάσταση βρίσκεται και η Ελβετία. Δηλαδή η Ελβετία μοιάζει περίπου με, τη να έχει, βρίσκεται στην ίδια θέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πιστεύω ότι θα εξελιχθεί η θέση της Ελβετίας ακριβώς επειδή αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών που πιέζουν για τη δέουσα επιμέλεια και βέβαια θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι και η τελική θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αν ουσιαστικά συμμετάσχει. Για τον Καναδά, για την Ιαπωνία είναι αβέβαιο ποια είναι η θέση του και σα ανέφερα μόνο λίγε από τι χώρε. Θα διαφωνήσω με εκείνον τον ομιλητή, ο οποίο είπε ότι τώρα ολοκληρώθηκε η συνθήκη. Αντιθέτω, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρώτο προσχέδιο, το οποίο διανεμήθη στι αντιπροσωπείε και συζητείται ακόμα. Είναι ανοιχτό το ερώτημα του κατά πόσον θα δοθεί και τι θα περιλαμβάνει μια διαπραγματευτική εντολή. Κατά την άποψή μας, θα ήταν σκόπιμο να δοθεί διαπραγματευτική εντολή στη νέα ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει εξελίξεις και είναι σημαντικό να μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να απαντήσει στο ερώτημα εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να συμμετάσχει σε αυτή τη διαπραγμάτευση ή όχι και πώς. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα που θα απασχολήσει την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά εγώ δεν μπορώ να προκαταλάβω τι πρόκειται να κάνει η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι άλλο σημαντικό, το ανέφεραν και πολλοί από, τους, από τα μέλη του Κοινοβουλίου, είναι το τι πρωτοβουλίες αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο εσωτερικό της. Γιατί γνωρίζουμε ότι το, το Μάρτιο μάλλον του 2018 είχαμε κατευθυντήριες οδηγίες ε, και ξεκίνησε και μια μελέτη από τη Γενική Διεύθυνση ε, Δικαιοσύνη για τη δυνατότητα να υπάρξει μια εγκάρση νομική πρωτοβουλία, νομικό κείμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ε, δεύτερη επιμέλεια. Όπω σα είπα, έχουμε επαφέ με τρίτε χώρε στην Γενέβη. Όμως όλα εξαρτώνται από τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλε. Μπορεί επί της αρχής να συμφωνούμε στη δέουσα επιμέλεια, αλλά είναι κάτι διαφορετικό το να το αναλάβουμε ω νομική υποχρέωση. Και συμφωνώ επίσης και με την ε, κυρία Αρένα, δεν είναι πυρηνική φυσική, πρέπει κανείς να λάβει μια απόφαση. Ποια είναι η διαπραγματευτική εντολή που δίνει στην Κομισιόν και μέχρι πού φτάνει αυτή. Επίση, πιστεύω ότι αυτό θα έχει σημασία και για τη μελλοντική εξέλιξη του ευρωπαϊκού δικαίου σε σχέση με τα ζητήματα δέουσα επιμέλεια. Και ευελπιστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, κατευθύνει εκείνο τι εξελίξει σε αυτόν τον τομέα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. κατευθύνοντα αντιστοιχώ και τη θέση που θα λάβουμε στο διεθνέ επίπεδο. Φαντάζομαι όλοι γνωρίζετε ότι όταν το Συμβουλίο Υπουργών Εξωτερικών συνέρχεται με την ε, μορφή ε, διεθνού εμπορίου, με τη σύνθεση διεθνού εμπορίου, κάτι που θα συμβεί σε λιγότερο από 7-8 μέρες, ε, τίθεται το ζήτημα υπό τα διάφορα για την συμπεριφορά των επιχειρήσεων, αλλά αυτό οδηγεί πάντα σε μια πολύ σύντομη συζήτηση στο περιθώριο του Συμβουλίου. Συμφωνώ με εκείνους που είπαν ότι αν φροντίσουμε τα του οίκου μας θα έχουμε καλύτερη διαπραγματευτική θέση και στη Γενέβη. Πράγματι και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το φροντίσουμε ανεξαρτήτως και προτού λάβουμε οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση με τις διαπραγματευτικές εντολές. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα έχουν απαντηθεί απευθείας ή έμεσα όλες οι ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Αν κάτι έχω ξεχάσει, θυμίστε το μου παρακαλώ. Α, ναι, για τα συμπεράσματα των ε, εισηγητών και τις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν και διαπεριφερειακές διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά τις προτάσεις διατύπωσης χωρίς ε, διαπραγματεύσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι σε θέση να σχολιάσει πέρα από αυτά που έχει ήδη σχολιάσει κατά τη διάρκεια της Συνόδου στις παρουσιάσεις. Τα υπόλοιπα εξαρτώνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά είμαι σίγουρος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πιέσει για τη δέουσα επιμέλεια. Και να ξέρετε ότι δεν είμαι εγώ που πρέπει να πείσετε ότι λειτουργεί η δέουσα επιμέλεια, αλλά τους νέους επιτρόπους. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρουμε, έχουμε συνεργαστεί μαζί σας και ξέρουμε ότι γνωρίζετε πολλά για τη δέουσα επιμέλεια εσείς. Έχετε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς έχουμε ψηφίσει πολλά ψηφίσματα. Οπότε δεν χρειάζεται να περιμένετε περισσότερο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ακολουθήσει το ψήφισμά μας. Έχουμε δουλέψει πολύ πάνω σε αυτά. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας εδώ και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Λοιπόν, τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη της ε, Υποπιτροπής μας Επόμενη συνεδρίαση 2 Δεκεμβρίου 3 με 6 και 30 μετά μεσημβρίες και 3 Δεκεμβρίου 9 με 12 και 30 και 14 και 30 με 18 και 30. Καλό βράδυ σε όλους. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίασή μας.